Ja, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Ausschusssitzung. Wie ich heute Morgen angekündigt Όπως έχω την ευχαρίστηση να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας την Πατρίτσια Εσπινόζα Καντελάνο, η οποία είναι Υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού. η οποία είναι πρόεδρος της COP16 στο Κανκούν. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Έχουμε επίσης εδώ και τη, τον πρόεδρο Σάντα Φουέντες, τον πρέσβη, συγγνώμη, του Μεξικού Σάντα Φουέντες. Την, την πρέσβη. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Μεξικό. Ο Ρικάρτο Κόρδες είναι επίσης εδώ. Καλώς όρισες. Κυρία Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος που πραγματικά παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, κινητήρια δύναμη για την προστασία του περιβάλλοντος. Σας καλωσορίζει εδώ Είχαμε μια συζήτηση σήμερα το πρωί για το ποσοστό των 20%, αν θα το ξεπεράσουμε, αν θα ανέβουμε, αν θα το πετύχουμε. Ε, Βεβαίω εδώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το 20%, 30% και βεβαίως ε, υπάρχουν αντιπροσωπείς από όλες τις πολιτικές ε, δυνάμεις και πολλοί από εμά ε, περιμένουν να υπάρξει επιτυχία σε αυτό το κάψι 16 και βεβαίως όπως όλοι οι συμμετέχοντες περιμένουμε μετά την ΚΑΠ 15 να προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα στην Κανκούν για το μέλλον. Θα σταματήσω όμως εδώ τα σχόλιά μου, τα εισαγωγικά μου λόγια, γιατί στις 4 ε, παρατέταρτο έχουμε τον κύριο Έτιγκερ, τον Επίτροπο, μέχρι τις 4.30 μπορεί να μείνει μαζί μας και θα μας μιλήσει για την ε, πολιτική του όσον αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την καταστροφή στην Ιαπωνία. Και βεβαίως μπορείτε να μιλήσετε Ισπανικά. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μένα είναι τιμή να μπορώ να παρευρίσκομαι εδώ σήμερα με όλους εσάς, ενώπιόν σας. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι το Μεξικό τιμά βαθιά τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά στο πλαίσιο αυτό η σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και θα ήθελα επίσης να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή για να σας εκφράσω όσα είπα σήμερα το πρωί στο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι δηλαδή το Μεξικό επιθυμεί να διατηρήσει μία θεσμική και ένα μόνιμο σχέση και ένα μόνιμο διάλογο για οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να ενδιαφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά τις διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αδράτω την ευκαιρία για να σας κοινοποιήσω πόσο μεγάλη ικανοποίηση ήταν για το Μεξικό να μπορέσει να οδηγήσει σε καλό λιμένα τις διαπραγματεύσεις ε, του Κανκούν και να τονίσω το ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαδικασία. Αν μου επιτρέπετε, θα περάσω κατευθείαν στην ουσία του ζητήματος, ε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε και κάποια ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω ορισμένα εισαγωγικά σχόλια. Καταρχήν, Το Μεξικό αποτελεί μια χώρα πεπισμένη ότι η επίλυση της κλιματικής αλλαγής όπως και των μεγάλων παγκόσμιων προβλημάτων έγκυται στη διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών βημάτων που οικοδομούμε εδώ και τόσο καιρό με τόσο πολλή δουλειά. Πιστεύουμε στον πολυμερισμό, εργαζόμαστε σε αυτά τα βήματα, σε αυτά τα φόρα για να βρούμε κοινέ λύσεις σε κοινά προβλήματα. Όπως γνωρίζετε, η προετοιμασία της συνδιάσκεψης ε, του Κανκούν και η διαιοθέτηση των συμφωνιών ήταν ε, πολύπλοκες ε, όχι μόνο λόγω των, τεχνικών δυσκολιών του ζητήματος αλλά και λόγω της μεγάλης ε, δυσπιστίας που εμπόδισε να, να μεταφραστούν έτη διαπραγματεύσεων σε συγκεκριμένες συμφωνίες. Και αυτή η δυσπιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνη προερχόταν από το ότι πολλές κυβερνήσεις είχαν εντοπίσει την αναγκαιότητα ενεργειακού εφοδιασμού για την εξάλληψη της ε, ανέχειας. Είχαν ε, υιοθετήσει πάρα πολύ άκαμπτες θέσεις που δεν επέτρεπαν ε, να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν γίνει σεβαστοί, σεβαστές και οι δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί. Στο Διεθνές στη διεθνή σκηνή θέλουμε να υπερισχύσει το παγκόσμιο συμφέρον και όλα τα κράτη-μέρη της σύμβασης και οι πρωταγωνιστές ε, της ε, κοινωνία. Στο θέμα αυτό θέλαμε να έχουμε ένα ρεαλιστικό σενάριο που να μας ε, επιτρέψει να προχωρήσουμε σταδιακά στην επίτευξη των στόχων μας και Σιγά σιγά αυξάνουμε και τα επίπεδα φιλοδοξίας μας και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να αυξήσει αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας. Βεβαίως οι συμφωνίες του Κανκούν δεν είναι η οριστική λύση για την απάντηση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και πιστεύω ότι οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν Δηλαδή ότι υπήρχε ένας μόνος τρόπος για την επίτευξη μιας καθολικής λύσης του προβλήματος ε, της κλιματικής αλλαγής, ίσως να είχαν προκαλέσει μια λανθασμένη αντίληψη στην κοινή γνώμη και στη διεθνή κοινότητα, κατά την άποψή μου. Όμως, ε, παρόλα αυτά, οι συμφωνίες του Κανκούν μας δείχνουν ε, ότι ο καθολικός διάλογος και η συμμετοχή στις πολυμερείς διαδικασίες καλή διπίστη μας επιτρέπουν να αναλάβουμε δράση ενωμένη για ένα καλύτερο μέλλον ε, για τους λαούς μας τι μας αναλογεί να πράξουμε τώρα, μας αναλογεί να ενισχύσουμε τις προσπαθίες μας έτσι ώστε να πετύχουμε ότι οι συμφωνίες που υθετήθηκαν στο Κανκούν θα μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή. Και ποια είναι τα κεντρικά στοιχεία αυτών των συμφωνιών της διάσκεψης των Κανκούν. Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω το στοιχείο της ε, σταδιακής ε, πρόοδου, χωρίς να ξεχνάμε ότι η διεθνή κοινότητα φυσικά πρέπει να δράσει όσο το δυνατόν ταχύτερα για να αποφύγουμε μεγαλύτερο κόστος ε, των συνεπειών ε, των κλιματικών αλλαγών. Οι συμφωνίες του Κανκούν ε, παγιώνουν μια σταδιακή εστίαση για τη μείωση των εκπομπών και των περιοδικών αναθεωρήσεων που θα μας επιτρέψουν να ε, μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου σε ό,τι αφορά την άνοδο της ε, θερμοκρασίας στον πλανήτη. Όλοι στο πλαίσιο των κοινών τους, αλλά διαφοροποιημένων ε, ευθυνών τους και ικανοτήτων τους δέχτηκαν να συνεισφέρουν στην, κοινωνική προσπά... στην καθολική προσπάθεια υπομορφή διαφάνειας και εδώ ε, η επιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπής της ε, θέσης στο να θέσει τους δύο βαθμούς ως μακροπρόθεσμο στόχο και στον επιμένει στο στόχο αυτό με σαφείς πρωταγωνιστές στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ε, που πολύ καιρό είχαν αποκλίνουσες απόψεις Ορισμένοι ήθελαν ε, να πετύχουν ένα πιο φιλόδοξο στόχο ε, κάτω των ε, δύο βαθμών Κελσίου, ενώ άλλοι δεν ήθελαν να αναλάβουν καμία δέσμευση σχετικά, όμως αυτή η συνεπής θέση, κάθε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κεντρικό στοιχείο για να καταλήξουμε στη συμφωνία, στη συνεννόηση. Ξέρουμε παρόλα αυτά ότι ακόμη και ο στόχος αυτός μπορεί να οδηγήσει σε ε, εξαιρετικές περιπτώσεις ε, σε πολλές χώρες. Γι' αυτό ε, βάσει των επιστημονικών στοιχείων που θα έχουμε στη διάθεσή μας θα προβαίνουμε σε διαρκείς αναθεωρήσεις ε, έτσι ώστε αυτή η θερμοκρασία να διατηρείται κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Υπάρχουν ε, κάποια νησιωτικά κράτη, ε, κάποια αναπτυσσόμενα κράτη που θα φυγούν πολύ σοβαρά αν δεν κατορθώσουμε να πάμε σε ένα στόχο πέρα των δύο βαθμών. Κελσίου. Όμως αυτή τη στιγμή πολιτικά δεν ήταν βιώσιμη μία συμφωνία που να θέτει ένα στόχο κατώτερο και κατορθώσαμε οι χώρες που συνεχίζουν να διατηρούν μια κάθετη θέση για την αναγκαιότητα να πάμε πιο πέρα, να συνοδεύσουν ε, αυτό το πακέτο αποφάσεων, ε, να το θεωρήσουν ως ένα συνενετικό πακέτο. παρόλα αυτά, αν ε, δεν επιτευχθεί ο τελικός ε, στόχος, ε, παρόλα αυτά θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε διάφορους πυλώνες που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Επίσης είχαμε και μία δέσμη μέτρων για το μετριασμό τόσο για τις χώρες του παραρτήματος 1 όπως και για τις αναπτυσσόμενες χώρες όπου Εκεί μιλάμε και για συμβασμό αλλά και για εθνικέ δράσεις μετριασμού, για εκούσιες δράσεις. Όμως παρόλα αυτά αν μετατραπούν σε δεσμεύσεις θα είναι κάτι πολύ θετικό και αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να αναθεωρηθούν, θέλουμε να τους αναθεωρήσουμε υπό το φως και της ε, ε, προόδου που έχει σημειωθεί σε επιστημονικό επίπεδο και σε τεχνολογικό επίπεδο για να μπορέσουμε τελικά να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι οι δεσμεύσεις και οι δράσεις μετριασμού των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών που κατορθώσαμε να εισαγάγουμε τις συμφωνίες του Κανκούν ουσιαστικά σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες από αυτές που προβλέπονταν στο αρχικό πρωτόκολλο του Κιώτου. Οι αναπτυγμένες χώρες ανακοίνωσαν ε, τα ε, στόχους μείωσης εκπομπών τους και φυσικά με ευρία νομιμότητα και οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, ανακοίνωσαν τους δικούς τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αυτή η αλλαγή προς μια συλλογική προσπάθεια ήταν θεμελιώδης για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα με ευρεία υποστήριξη. Ένα άλλο στοιχείο των συμφωνιών του Κανκούν που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξή. Ε, κατορθώνουμε να προσδιορίσουμε μια θεσμική αρχιτεκτονική στήριξη στον αναπτυσσόμενο κόσμο στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Όπω γνωρίζετε, συμπεριλαμβάνει το μηχανισμό μείωση των εκπομπών ε, λόγω της αποψήλωση ε, των δασών και της διάβρωσης του εδάφους Red Plus, όπως είναι γνωστό, Red Sea. Επίσης, συμπεριλαμβάνει την ε, δημιουργία πλαισίου προσαρμογής του Κανκούν που είναι πολύ πιο σχετικό όταν ε, βλέπουμε ε, τι συμβαίνει σε διάφορες περιοχές του κόσμου, τα κρέα καιρικά φαινόμενα. Πέρσι είχαμε τις περκαγιές στη Ρωσία, τις πλημμύρες στο Πακιστάν, τις ξηρασίες στην Αφρική, καύσονες εδώ στην Ευρώπη ή τις, πολλές, τις πολύ μεγάλες χιονοπτώσεις που είχαμε σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και στο Μεξικό. Είναι τμήμα της ζωής μας και αυτό. Έχουμε ε, τους, ε, τις πλημμύρες ε, που είναι αποτέλεσμα των τυφώνων. Έτσι λοιπόν ε, αυτό το πλαίσιο υποστήριξης για την προσαρμογή αποτελεί ένα ζωτικό εργαλείο κυρίως για τις πιο μικρές χώρες που φύγονται τα μάλα από την κλιματική αλλαγή και δεν έχουν την ικανότητα να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες και ούτε υπάρχουν ακόμη τα τεχνικά ή τα οικονομικά μέσα στον κόσμο σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας για να στηρίξουμε συγκεκριμένα αυτές τις χώρες στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτό το πλαίσιο προσαρμογής συνοδεύεται επίσης από τη δημιουργία ενός ε, τεχνολογικού μηχανισμού που θα επιτρέψει τη δημιουργία δικτύων και περιφερειακών ε, ή εθνικών ε, κέντρων τεχνολογίας όπως και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη δημιουργία ικανοτήτων. Είναι γεγονός ότι όσοι επένδυαν στην ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών απαιτούν οι τεχνολογίες τους να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή θέλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύ η ατζέντα σε αυτό το τομέα και αυτός ήταν και ένας τρόπος να δημιουργηθούν τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου να συνεχίζουν να γίνονται αυτές οι επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ταυτόχρονα να συνεχίζουν να ωφελούνται οι κοινωνίες των χωρών όπου εφαρμόζονται οι τεχνολογίες αυτές. Δηλαδή στην πραγματικότητα εδώ επιζητούμε να δημιουργήσουμε ένα φαυλοκύκλο που θα έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια βρία στρατηγική για την ε, κλιματική αλλαγή και στις ε, φτωχές, στις μικρές, στις αναπτυσσόμενες χώρες που αποτελούν μια αγορά για τις τεχνολογίες αυτές και μέσω των μηχανισμών που έχουν το στόχο να διευκολύνουν αυτές τις τεχνολογίες, την πρόσβαση μάλλον, σε αυτές τις τεχνολογίες, Επίσης, επιτρέπουν στις χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερες δεσμεύσεις από ό,τι κανονικά θα μπορούσαν να αναλάβουν, γιατί δεν θα είχαν αυτή τη στήριξη. Συμφωνήσαμε επίσης σε κάτι πολύ σημαντικό για ε, το κλιματικό καθεστώς του μέλλοντος, τη δημιουργία του Πράσινου Ταμείου για την κλιματική αλλαγή, που έχει το στόχο να προβλέπει χρηματοδότηση, να εξασφαλίζει χρηματοδότηση για τα προγράμματα στι αναπτυσσόμενε χώρε. Και φυσικά αναγνωρίστηκε και το εξή. Προσφορά χρηματοδότησης ε, στο πλαίσιο των ε, κονδυλίων ε, ταχείας εκκίνησης που μπορούν να ε, μεταφερθούν από τις αναπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες στην περίοδο 2010-2012. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ότι στη συνδιάσκεψη του Κανκούν ε, υπήρξε ένα στοιχείο που κατά την άποψή μου ήταν πολύ σημαντικό για τον εμπλουτισμό των συζητήσεών μας και στη συνεισφορά σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια, η συμμετοχή δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών, ε, του ιδιωτικού τομέα, των ακαδημαϊκών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και των νομοθετών. Θα ήθελα να σας πω ότι το Μεξικό πρότεινε επισήμω να αναγνωριστούν οι νομοθέτες στο πλαίσιο της σύμβασης ως ε, μια ειδική ομάδα ενδιαφέροντος. Γιατί? Εγώ δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω εδώ πόσο σημαντικό είναι το δικό σας έργο για να επιτρέψετε να γίνουν σεβαστοί οι στόχοι των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν οι κυβερνήσει μας. Δυστυχώ στο Κανκούν δεν υπήρχε συνένεση για να μπορέσουμε να θετήσουμε αυτή την τροποποίηση, αλλά ελπίζουμε και ελπίζουμε να μας βοηθήσετε για να διευρυνθεί αυτή η συμμετοχή προς τους νομοθέτες των διάφορων χωρών Θα πρέπει να δούμε βέβαια με ποιο τρόπο θα γίνει. Όμως πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι νομοθετικές αρμοδιότητες αποτελούν τμήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των κρατών. Τι κάνουμε εμείς ε, τώρα ως Προεδρία της διάσκεψης των μερών. Προσπαθούμε από κοινού με την Υπουργό Εξωτερικών Σχέσεων της Νοτιοαφρικής που διορίστηκε από τον πρόεδρο για να ε, προεδρεύσει της διάσκεψης του Ντουρμπάν να καθορίσουμε το πρόγραμμα που θα θέσουμε σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του έτους. Οι προοπτικές ε, προς τη διάσκεψη του Ντουρμπάν είναι μικτές δεν ε, θέλω να είμαι ούτε υπερβολικά αισιόδοξη, ούτε υπερβολικά απεσιόδοξη. Έχουμε το πλεονέκτημα, σε αντίθεση με ό,τι έγινε με το Κανκούν. Τώρα έχουμε μια πολύ σαφή στρατηγική για το τι πρέπει να κάνουμε, μια να θέσουμε σε εφαρμογή ένα παγκόσμιο καθεστώ κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα όμως Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που δεν καν έχουμε ξεκινήσει να τα συζητάμε. Το θέμα της χρηματοδότησης, παραδείγματο χάρη. το θέμα αυτό η συζήτηση επικεντρώθηκε μέχρι τώρα στο αν θα δημιουργούταν ή όχι ένα νέο ταμείο. Τώρα όμως πρέπει να περάσουμε στη συζήτηση για το πώς θα λειτουργήσει το ταμείο αυτό, από πού θα προέλθουν οι πόροι. Κατά την άποψη του Μεξικού, εμείς ε, είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο θα υπάρξει δημόσια χρηματοδότηση, αλλά και ένα τμήμα των κονδυλίων που θα ενεργοποιηθούν θα πρέπει να προελθούν και από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί μιλάμε για ένα ελάχιστο στόχο. 100 ε, δις ε, δολάρια το χρόνο μέχρι το 2020. Και πρέπει να πούμε ότι η αγορά σε ό,τι αφορά τις ε, υπηρεσίες ε, στο περιβαλλοντικό τομέα, ορισμένοι του υπολογίζουν ως 500 δις ε, το χρόνο. Υπάρχει εδώ ένα σημαντικό επίπεδο επιχειρήσεων που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, όμως ε, ξέρετε ότι πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται στι λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε ταχύτατα. Και τα θα μπορούσα να πω και για το μηχανισμό Red Sin, για την Επιτροπή Προσαρμογής. Ε, τώρα πρέπει να αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε επί των λεπτομεριών. Και σε αυτή τη διαδικασία μας είναι απαραίτητη όλη η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υλοποιεί ένα σημαντικό έργο. Σας είπα ήδη πώς συνεισφέρει η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση ε, γεφυρών μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Επίσης, ε, συνεισφέρει στο να μην βλέπουμε αυτό το θέμα ως ένα ζήτημα γιατί πρόκειται για ένα θέμα και είναι ενδιαφέροντος για την ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν, κατά την άποψή μου, ενέχει και τη δυναμική επαναπροσδιορισμού των γενικών θεωριών για την αναπτυξιακή βοήθεια. Εμείς όταν μιλάμε για αναπτυξιακή βοήθεια σκεπτόμαστε τη δράση μιας χώρας που είναι πιο πλούσια και μπορεί να βοηθήσει μια χώρα που βρίσκεται σε πιο μειονεκτική θέση. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχοντας ε, αυτή τη στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, όχι μόνο βοηθούμε τις χώρες αυτές, αλλά δημιουργείται και ένα κοινό αγαθό που είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Σας επαναλαμβάνω για να κλείσω ότι το Μεξικό δεσμεύεται στο να συνεχίζει τις εργασίες στον τομέα αυτό. Σας ζητώ και πάλι την υποστήριξή σας τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και στις σχέσεις με τους λοιπούς ε, εταίρους της διεθνούς κοινότητας. Γιατί, επαναλαμβάνω, εδώ η προσπάθεια όλων είναι απαραίτητη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι κάνατε εξαιρετική δουλειά και στο Κανκούν. Ίσως δεν θα σας ευχαριστήσουν όλοι. Εγώ μιλώ εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής και μετά Κανκούν ήμασταν όλοι ευτυχείς. Το θέμα είναι τώρα πρέπει οι δεσμεύσεις αυτές να αρχίσουν να υλοποιούνται και να προσθεθούν βεβαίως και κάποια επιπλέον στοιχεία όσον αφορά ένα συνολικό πακέτο συμφωνίας για το κλίμα. Ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σας. Ο κάθε ομιλητής θα πρέπει όμως τώρα να πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Έχετε σχόλια, έχετε ερωτήσεις για ένα λεπτό. Ο κύριος Φλόρεντς, παρακαλώ πολύ ένα λεπτό. Δεν είναι εύκολο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό. Και βεβαίως ε, δεν ήταν εύκολο κανείς να συνεχίσει την Κοπενχάγη. Είδαμε όμως τι συνέβη σήμερα στην Ιαπωνία και στο Ντουρμπάν. Θα πρέπει βεβαίως να περάσουμε στην επόμενη φάση των αποφάσεών μας. Τι την εντύπωση έχω. Το θέμα της αποψήλωσης επίσης είναι ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα γιατί υπάρχουν εδώ θέματα που αφορούν ε, και την οικονομία, τεράστια θέματα. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι το θέμα της διπλωματικής υπηρεσίας με θέμα το κλίμα. Είναι κάτι που επιθυμούμε να ενισχυθεί στην Ευρώπη. Παρακολουθούμε ότι πολλές χώρες έχουν διμερείς ε, διαπραγματεύσεις, συμφωνίες αλλά σε πολυμερές επίπεδο θεωρούμε ότι η Ευρώπη έχει δυνατότητα να κάνει παραπάνω. Τι λέτε γι' αυτό. Thank you, Yes. Yeah. Minister, I also... Ευχαριστώ. Και εγώ έχω γράψει ήδη κάποια σχέδια επένων για σας, αλλά θα τα πω γιατί δεν έχω χρόνο. Θα περάσω κατευθείαν σε ερωτήσεις. Τι θα γίνει με το πρωτόκολλο του Κιώτο. Θα έχουμε μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων. Πιστεύετε, είναι σόφρον η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει στεναρή, α, ανάλογη προς τις δεσμεύσεις της πρώτης περίοδου. Επίσης, το θέμα του μετριασμού των κλιματικών αλλαγών δεν το έχουμε ακόμα ελέγξει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι άλλοι σημαντικοί εταίροι που δεν έχουν μετακινηθεί ακόμα θα αλλάξουν στάση στον Τέρμπαν. Τι θα γίνει στον Τέρμπαν, αν δεν υπάρξει κανένα μέτρο για το μετριασμό. Τρίτη ερώτηση. Ποια είναι η συμβουλή σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνουμε από τώρα μέχρι τον Τέρμπαν για να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Πρώτη ήταν το ΕΛΚΑ, ε, μετά ήταν οι σοσιαλιστές και τώρα είναι οι φιλελεύθεροι με τον Chris Ντέιβις. Εμείς συζητάμε αν θα πρέπει να αυξήσουμε τους στόχους μείωσης του διοξείδου του άνθρακα η δέσμευση ε, στο παρελθόν είναι ότι θα το κάνουμε μόνο αν υπήρχε μια δεσμευτική διεθνή συμφωνία. Κοιτάζω τώρα προς το μέλλον. Δεν βλέπω προοπτικές να υπάρξει συμφωνία δεσμευτική που θα ικανοποιεί τις κυβερνήσεις που είναι απρόθυμες να προβούν σε μέτρα που εμείς θα θέλαμε, τουλάχιστον αυτήν την Επιτροπή, να λάβουμε. Ε, από το Κιώτο και μετά ε, πώς θα προχωρήσουμε. Ε, εσείς τι πιστεύετε, ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα α, δεσμευτικής συμφωνίας κάποια στιγμή, στο εγγύς όμως μέλλον. Χάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, Υπουργό και να την επενέσω. Η ερώτησή μου συνδέεται με αυτά που είπε ο Chris Davis. Οι χώρες ε, ήταν πολύ σημαντικό να συμφωνήσουν οι χώρες στο Κανκούν για αυτό το στόχο του δύο, των δύο βαθμών Κελσίου. Αλλά οι δεσμεύσεις για τις εκπομπές ε, στην ε, Κοπενχάγη που επισημοποιήθηκαν στην, ε, στο Κανκούν, στην πραγματικότητα δεν συνάδουν με το στόχο του, των δύο βαθμών, όπως είπατε κι εσείς. Ποια είναι λοιπόν η συμβουλή σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να κάνουμε εμείς για να προωθήσουμε μια συμφωνία, για να διευκολύνουμε μια συμφωνία. Και οι δικοί μας στόχοι για τη μείωση των εκπομπών ε, συνάδουν με το στόχο ε, της μείωσης ε, της θερμοκρασίας των δύο βαθμών από τους αριστερούς τώρα. Η κυρία Ντεμπρούν. μετά από τη Συμφωνία του Κανκούν, ένα σημαντικό πράγμα είναι οι καταιγιστικές προθεσμίες ούτω ώστε τα μέρη να υποβάλουν πληροφορίε και απόψει για μια σειρά από θέματα. Διερωτώ με, αν θα μπορούσατε να μου δώσετε τι απόψει σα για αυτά τα έγγραφα και τι προτάσει που υποβλήθηκαν μέχρι στιγμή. Κάποιου μηχανισμού που να μην βασίζονται στην αγορά, α πούμε. Ε, μπορείτε να μου του σχολιάσετε. και κάποια θέματα όπως οι πληροφορίες από τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες για, τον, για τις δράσεις για τον μετριασμό, ας πούμε, που δεν συνοδεύονται από προθεσμίες. Μπορείτε να μου τις σχολιάσετε. Στις 14 και 15 Μαρτίου θα συζητήσουμε για, θα συζητούσαμε μάλλον για το πράσινο αυτό ταμείο, αλλά να βγάλετε αυτή η συνάντηση. Γιατί? Όλοι ε, σέβονται το χρόνο τους. Ε, σας, σας ε, μέσα σε ένα λεπτό μίλησαν όλοι οι προηγούμενοι. Σας, σας δίνω πέντε λεφτά. Είναι εντυπωσιακό το ότι μπορεί να πει κανεί μέσα σε πέντε λεφτά. Σας θαυμάζω που θέτετε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσε πολλέ ερωτήσεις για την αποψήλωση των δασών. Συμφωνώ πλήρω. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό. Είναι η τρίτη πηγή εκπομπών παγκόσμια. Πρέπει να προσέξουμε. Θα υπάρξουν και πολλά κοινωνικά ωφέλη σε χώρες όπου υπάρξουν προγράμματα αναδάσωσης. Με βάση την εμπειρία λοιπόν που έχουμε, από τα βήματα που έχουμε ολοκληρώσει μέχρι στιγμής, να ένας τομέας όπου θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κάτι το απτό, να υπάρξει κάτι το απτό στον Τέρμπαν. Τώρα, κάτι άλλο που συνδέεται με αυτό. Τι θα γίνει με το πρωτόκολλο του Κιώτο. Πιστεύω ότι καθαρές συμφωνίες για μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων ή δεσμευτική περίοδο δεν είναι η πραγματική λύση. Δεν είναι η πανάκια. Δεν σαν θέλουμε να πούμε ας εγκρίνουμε, ας πούμε, ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση της στόχιας και θεωρούμε ότι το ψήφισμα από μόνο του θα σταματήσει τη φτώχεια. Φυσικά πρέπει να σκεφτούμε τι είδους δεσμεύσεις και τι είδους καθεστώς θέλουμε να δημιουργήσουμε μετά το 2012. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι οι δεσμεύσεις που έθεσαν επιτάβητος οι χώρες ξεπερνούν το 2012. Και το πρωτόκολλο του Κιώτου του Κιώτο παραμένει ενισχύ μετά το 2012. Ούτως ή άλλως δεν έχει ημερομηνία εκπνοής. Οι στόχοι που είχαν τεθεί για την πρώτη περίοδο δεσμεύσεων θα εξακολουθήσουν, υποτίθεται, να ισχύουν και μετά το 2012. Γιατί, Γιατί δεν πρόκειται να τους υλοποιήσουμε το 2012. Το πρωτόκολλο Δηλαδή η νομική βάση επί της οποίας οι χώρες υποχρεούνται να προβούν σε αυτές τις δράσεις για να καταπολεμήσουν την ε, κλιματική λαγή, όλα αυτά παραμένουν ισχύ. Το πρωτόκολλο ισχύει λοιπόν. Θα πρέπει να δούμε τώρα τα μέσα που θα εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας για όλους. Αυτό συνδέεται πολύ με την εφαρμογή τη συμφωνία του Κανκούν. Αν αρχίσει να λειτουργεί αυτό το ταμείο, το πράσινο ταμείο, θα μπορέσουμε να ζητήσουμε περισσότερες δεσμεύσεις από τι αναπτυσσόμενε χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενε οικονομίες. Φυσικά, όπως ξέρετε, το Μεξικό στον αναπτυσσόμενο χώρο ήταν μία από αυτούς που ήθελαν να αναλάβουν περισσότερες δεσμεύσει. Γιατί, είναι η πραγματικότητα, μας επηρεάζει όλους. Ε, δημιουργεί και οικονομικό κόστος, αλλά πλήττει και τις ανθρώπινες ζωές. Ε, μας βαραίνει όλους. Επομένως, έχουμε συμφέρον να κάνουμε κάτι. Και δεσμευτήκαμε γι' αυτό. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας λοιπόν. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε λοιπόν καταρχάς την εντολή του Κανκούν, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε τα μέσα που θα επιτρέψει στις χώρες να περάσουν σε περισσότερες δεσμεύσεις. Δεν επιταγεί εν λευκό που τη δίνουμε στις αντισώμενες χώρες για να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι. Τους δίνουμε αυτά λεφτά για προγράμματα καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε το συντομότερο δυνατόν κάποιες διαδικασίες ούτως ώστε να φτάσουμε σε κάποιες νέες τεχνολογίες και αυτή την πρόσβαση να την έχουν πολλές χώρες, ώστε να τον περισσότερες. Μόνο έτσι θα είναι προσιτές οι τεχνολογίες αυτές, μόνο έτσι θα έχουμε τα κίνητρα για να υπάρξουν περαιτέρω επενδύσεις και είναι ο μόνος τρόπος που οι αντισώμενες χώρες θα είναι σε θέση να καταβάλουν και αυτές τις προσπάθειες στο παιχνίδι αυτό. Σημερίζουμε την άποψη ότι είναι σαφές τι θα γίνει με την τελική απόφαση για το μέλλον του καθεστώτος μετά το 2012, όταν τελειώσει η πρώτη περίοδος σωσμεύσεων. Εδώ μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δούμε σε ποιο πολιτικό επίπεδο θα λάβουμε τις απόψει. Πρέπει να λυθούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Είναι τεχνικό το θέμα, ναι, αλλά χρειαζόμαστε πολιτικές αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να συνεργαστείτε εσεί. όλες οι κυβέρνησεις δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα τελικό σχόλιο για τη μεταβατική αυτή επιτροπή. Εμείς θέλαμε να σεβαστούμε την προθεσμία του Κανκούν, αλλά την αναβάλαμε γιατί υπήρχε μεγάλη αντίθεση από τις ασιατικέ χώρες, τη ΑΖΕΑΝ. Δεν, δεν θέλανε, γιατί δεν συμφωνούσαν στο ποιο θα εκπροσωπήσει τις χώρες αυτές σε αυτή τη μεταβατική επιτροπή. Αν έχετε λοιπόν φίλους στις χώρες ΑΖΕΑΝ, ε, να, ένα τρόπο για να μα βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε στις Βρυξέλλες. και που αφιερώσατε αυτό το χρόνο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, για τις εξηγήσεις σας. Ελπίζω να τα καταφέρουμε στον Τέρμπαν. Εμείς θα είμαστε παρόντες. Και έχετε προσκαλέσει και τους νομοθέτες. Όχι δηλαδή μόνο κυβερνήσεις, αλλά και νομοθέτες, την κοινωνία των πολιτών, δημάρχους, τοπικές αρχές κτλ. Όλες, όλοι οι φορείς αυτοί χρειάζονται ούτως ώστε να έχουμε μια ευρεία προσέγγιση για τον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Okay, der Kommissar schon da. Uh, Dann, äh,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 Ich habe Sie gesucht draußen. Entschuldigung, da ich, Sie haben die Listen rausgekleidet, dann durch <laughs> hochgekleidet. okay. Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να χαιρετήσω τον Επίτροπο Γκίντερ Χέτιγκερ για ενέργεια, αρμόδιο για ενέργεια. Είσαστε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας ε, και βεβαίως τα γεγονότα στην Ιαπωνία μας έχουν ε, εξαιρετικά συγκινήσει και σοκάρει. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που μπορέσατε να βρείτε χρόνο και για μας. Ξέρω ότι ε, χτες ήσασταν στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Μέχρι τις 4.30 θα είστε εδώ μαζί μας και θα μας ενημερώσετε για αυτά τα οποία έχουν ε, γίνει. Και βεβαίως πρόκειται για μια χώρα, η Ιαπωνία, με εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία. Όλοι σήμερα λένε ότι όλα αυτά μπορεί να μας αφορούν και εμάς. Αλλά δεν θέλω να χάσουμε κι άλλο χρόνο, κύριε Επίτροπε. Υπάρχουν ε, πολλά που πρέπει να μας πείτε και σύμφωνα με τον χρόνο που έχουμε, ενδεχομένως να απαντήσετε και στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Κύριε Κυρίε Κυρίες και κύριοι, βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, βεβαίως με μεγάλη συγκίνηση κοιτάμε τις εικόνες από την Ιαπωνία και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος αυτής της τραγικής και πολύ μεγάλης καταστροφής θα συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα όλα αυτά δεν έχουν τελειώσει. Πριν από πέντε μέρες ακούσαμε ότι υπάρχει ένα σεισμό. Στην αρχή μας είπαν ότι ήταν 8,9 ρίχτερ, κατόπιν 9, 9,1. Κατόπιν είδαμε ότι υπήρξε μια μετακίνηση κατά δύο μέτρα της ε, ε, πλάκας που βρίσκεται κάτω από την Ιαπωνία. Κατόπιν ε, Άλλοι σεισμοί ακολούθησαν και το τσουνάμι, 10 μέτρα, 15 μέτρα. Τα ρεύματα που αναπτύχθηκαν στην περιοχή οδήγησαν σε διαφορετικές ε, μετατοπίσεις και σαν αποτέλεσμα αυτού Διακόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα, σταμάτησε η λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων και την ίδια ώρα, και αυτό ήταν και το πιο δυσάρεστο και επικίνδυνο, οι ε, μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται στους αντιδραστήρες για την ψήξη των συστημάτων. Ξέρετε τι έγινε στο Τσέρνομπιλ και πώς στην κλίμακα αυτών των καταστροφών αξιολογείται ο κίνδυνος. Εκεί ήταν 7 ε, στο Τσέρνομπιλ. Εχθές οι Ιάπωνες το αξιολόγησαν σε 5. Οι Γάλλοι ειδικοί θεωρούν ότι έχουμε φτάσει στο 6 σήμερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε στο 6 σήμερα και στην πυρηνική αυτή εγκατάσταση με ε, τους αντιδραστήρες αυτούς ε, της δεκαετίας του 70 είναι οι περισσότεροι. Βεβαίως, σήμερα ξέρουμε ότι τουλάχιστον ένας από, του, ένα από τα κέλυφος των αντιδραστήρων έχει πειραχθεί, υπάρχουν διαρροές και βλέπουμε σήμερα ότι και εκτός ελέγχου βρίσκεται η κατάσταση στην εγκατάσταση αυτή, από ό,τι τουλάχιστον μας λένε οι Ιαπωνές εμπειρογνώμονες. Και βεβαίως το σύστημα ψήξης έχει σταματήσει να λειτουργεί. Προσπαθούν να φέρουν ε, νερό από έξω και σε περίπτωση που η νέα αυτή επεξεργασία λειτουργήσει, παρόλα αυτά, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η ψήξη δεν γίνεται ούτε στο βαθμό ούτε με την ταχύτητα ε, που θα έπρεπε. Υπάρχει σήμερα λοιπόν διαφορετικές πληροφορίες και οι διαφορετικές αυτές πληροφορίες φαίνεται να γίνονται όλο και πιο διαφορετικές. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των νέων που μαθαίνουμε από την κυβέρνηση, αυτών που ακούμε από τους ειδικού τους εμπειρογνώμονες. Και ξέρετε πόσο ακριβείς είναι οι άπονες σε επιστημονικά θέματα. Τις επόμενες ώρες είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε δυστυχώς και άλλα δυσάρεστα καταστροφικά νέα. Το επικίνδυνο είναι αυτή τη στιγμή οι επιπτώσεις επί της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Σήμερα ξέρετε ότι η μεγαλύτερη Μητρόπολη του κόσμου, ε, το Τόκιο, ε, στο οποίο δεν επικρατεί ακόμα πανικός. Στην ε, Γαλλία αντίθετα η Υπουργό Περιβάλλοντος στη Γαλλία έχει δώσει εντολή στους Γάλλους που ζουν στην Ιαπωνία να εγκαταλείψουν την Ιαπωνία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι σαν να μην ζει κανένας άλλος σε αυτό το νησί. Εν πάση περιπτώσει, η διάσταση του προβλήματος είναι σήμερα πολύ δύσκολο να ε, αντιμετωπιστεί με ορθό τρόπο. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό για την δική μας ε, βιομηχανική πολιτική. Εχθές είχαμε μια πολύ σοβαρή συνέντευξη και συζήτηση από 7 διαφορετικά κράτη, με εμπειρογνώμονες, με υπουργού και βεβαίως τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές για θέματα πυρηνικής ενέργειας ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ατομικής ε, ενέργειας ήταν επίσης παρόντες και οι κατασκευαστές, όπως η Αρεβά παραδείγματο χάρη στη Γαλλία, πυρηνικών μονάδων. Και αυτή η συνάντηση υψηλού επίπεδου ε, έδειξε ότι σε κάποια σημεία υπάρχουν κοινέ θέσεις και σε κάποια άλλα διαφορετικές. Πού υπάρχουν διαφορετικές απόψεις παραδείγματος χάρη, εάν στο μέλλον το energy mix θα συνεχίσει να είναι αυτό που είναι σήμερα ή αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετικούς προσανατολισμούς. Εδώ δεν υπήρχε συμφωνία σε αυτό το θέμα. Εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης και δεν είμαι ο μόνος. Καταλαβαίνετε ότι οι θέσεις πλέον δεν είναι απλώς πολιτικές. Εχθές η πλειοψηφία, αν θέλετε, υπήρχε μία δυσπιστία αν ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα ενέργειας είναι αρκετά ουδέτερος, αρκετά αμερόληπτος και δεν επηρεάζεται από τις δικές του προσωπικές απόψεις για το θέμα. Και τελικά είδαμε ότι παραδείγματος χάρη για την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες δεν φάνηκε να ζητείτε μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια. Για τη Γερμανία, όπως ξέρετε, για την ε, Ελβετία και την Αυστρία, τρεις χώρες που είναι γερμανόφωνες, φάνηκε πάλι μια διαφορετική άποψη. Τελικά πετύχαμε όμως και σε κάποια σημεία μια κοινή θέση. Όλοι θέλουν να υπάρξει έλεγχος της ασφάλειας των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων. Και εδώ και δύο χρόνια η οδηγία για την ασφάλεια των ε, ευρωπαϊκών πυρηνικών εγκαταστάσεων, η οποία άρχισε να μεταφέρεται στις εθνικές νομοθεσίες, θα πρέπει βεβαίως να αποτελέσει την βάση αυτού του πρώτου βήματος. Εχθές όλοι είπαν ότι οι 143 πυρηνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ευρώπη θα πρέπει να περάσουν από έναν έλεγχο αντίστασης, ένα stress test με στόχο να υπάρξει μια νέα αξιολόγηση των κινδύνων βάσει της εμπειρίας της πρόσφατης από την Ιαπωνία. Το ερώτημα είναι αν στην Ευρώπη υπάρχει κίνδυνος για μια τέτοια πλημμύρα, για ένα τσουνάμι, αν μπορεί να υπάρξουν παραδείγματο χάρη εγκλήματα στον κυβερνό χώρο, επιθέσεις τρομοκρατικές με αεροσκάφη ή άλλου είδους κίνδυνοι που να πλήξουν αυτές τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, αν είναι αρκετά ε, ασφαλής, αν μπορεί να υπάρξουν προβλήματα τεχνολογικά, τεχνικά, ηλεκτρικής ε, ενέργειας, τροφοδοσίας κτλ. κτλ, κτλ. Και εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες θα ασχοληθούμε με αυτά γενικά αν θέλετε πρότυπα και κριτήρια βάσει των οποίων θα πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι. Θα εξετάσουμε επίσης την τοποθεσία αυτών των εγκαταστάσεων, αν είναι σεισμογενείς οι περιοχές. Θα εξετάσουμε βεβαίως και την ηλικία τους, την τεχνολογία που συνεχίζει να χρησιμοποιείται, τις κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά τα πρότυπα, την τις βέλτιστες πρακτικές και το πώς με τον καλύτερο τρόπο μπορούν να διενεργηθούν αυτοί οι έλεγχοι, αυτά τα stress test. Το ερώτημα που κάναμε χτες είναι ποια είναι τα πρότυπα ασφαλείας των κρατών μελών. Γιατί δεν μπορεί οι έλεγχοι αυτοί να γίνουν με διαφορετικό τρόπο στο κάθε κράτος μέλος. Πρέπει να βρούμε τα αυστηρότερα πρότυπα κριτήρια, τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Η ασφάλεια στην Ευρώπη είναι κάτι που δεν το διαπραγματευόμαστε. Δεν έχω καμία συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αυτών των ελέγχων, αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα υπάρχουν έτοιμες οι προδιαγραφές για αυτά τα stress test. Και από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος του χρόνου, και βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί και από τις εμπειρογνωμοσύνες, από τους ειδικού που διαθέτουμε, να προχωρήσουμε αμέσως σε αυτούς τους ελέγχους αξιοπιστίας. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει μέχρι τον Ιούλιο να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Και ως το 2014 θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός, μια αξιολόγηση και εγώ το θεωρώ αυτό πολύ αργά. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας ανακοινώσω αμέσως ότι αμέσως μετά αυτά τα stress test που θα γίνουν στις πυρηνικές καταστάσεις θα ζητήσω την ανανέωση, την τροποποίηση στο πρώτο εξάμεινο του 2012 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, έτσι ώστε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό κείμενο που να θέτει τα νέα πρότυπα για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Και βεβαίως να φτάσουμε στα απαραίτητα συμπαράσματα. Η χτεσινή υψηλού επίπεδου συνεδρίαση θα συνεχίσει τον Απρίλιο, θα επαναληφθεί και βεβαίως το Συμβούλιο θα ασχοληθεί, το Συμβούλιο Ενέργειας θα ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες. Θέλω επίσης να σας πω ότι την πέμπτη της επόμενης εβδομάδας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα ασχοληθεί κυρίως με το θέμα του ευρώ, της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, θα έχει σαν θέμα στην ημερήσια διάταξη εν ώψη των γεγονότων της Ιαπωνίας και το θέμα που συζητούμε σήμερα. Υπάρχουν χώρες όπως η Τουρκία, η Ελβετία, η Ρωσία που φυσικά ενδιαφέρονται και πολύ ε, ορθά ο κύριος Σαρκοζή θέλει να βάλει το θέμα αυτό και στην ημερησία διάταξη του G20. Αυτό θα πρέπει βεβαίως να το θίξει η ευρωπαϊκή διπλωματία και στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που έχουμε με την Ινδία και την Κίνα. Αυτά είχα να σας πω σαν εισαγωγικά σχόλια. Είμαι στη διάθεσή σας Ξέρω βεβαίω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη μέση διάταξη στην διάθεσή μας, συγγνώμη, αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα στην για διάταξη. Είμαι όμως στη διάθεσή σας και με χαρά θα ακούσω και τις επικρίσεις σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για αυτή την παρουσίαση. Πρέπει να σας πω ότι κατά την άποψή μας η αντίδραση της Επιτροπής είναι πολύ γρήγορη, πολύ γρήγορη αντίδραση επόμενη πέμπτη, αλλά θεωρώ πραγματικά ότι τα γεγονότα απαιτούν ταχεία αντίδραση και βεβαίως το ερώτημα είναι εδώ όχι μόνο ποια είναι η θέση μας σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Με ρώτησαν εχθές και σήμερα τι μπορεί να κάνει ο Επίτροπος τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή για αυτά τα θέματα, ποια είναι η αρμοδιότητά τους, υπάρχει αρμοδιότητα και αν πρέπει να πάψει να ισχύει η συνθήκη Euratom η συνθήση Euratom ενδεχομένως θα μπορούσε να τροποποιηθεί. Εδώ όμως έχουμε ένα πολύ πιο επίγον θέμα και δύσκολο πώς θα απαντηθούν 20 ερωτήσεις σε 20 λεπτά. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει καταρχήν να επιλέξουμε για ένα λεπτό έναν ομιλητή από την κάθε πολιτική ομάδα. Ο Φλόρεντς, Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πολύ για την δράση σας. Η κρίση αυτή είναι γνωστή και η δική μας αντίδραση όσον αφορά τα θέματα του κλίματος. Θα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε πώς θα αντιδράσει η Επιτροπή και πώς βλέπει το θέμα της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Ε, ε, Σε ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είσαστε εδώ, λέει η κυρία Σκόκ. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία των δοκιμών αντοχής είναι θαυμάσια ιδέα. Εγώ συμμετείχα σε μια κυβέρνηση που αποφάσισε να κλείσει ε, ένα πυρηνικό εργοστάσιο που λειτουργούσε μια χαρά και να ξεκινήσει τη διάλυση άλλων αντιδραστήρων σε μια ε, διαδικασία διαδοχικής κατάργησης των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ε, αυτές οι, αυτά τα μέτρα, έτσι, τα βραχυπρόθεσμα, δεν έχουν νόημα. Θα πρέπει να έχουμε μακρόπνοα σχέδια που θα μας οδηγήσουν προς άλλες ενεργειακές πηγές. Αυτό δεν είναι το ερώτημα που πρέπει να μπει στη μέση διάταξη. Την επόμενη εβδομάδα, όταν συναντήσετε τους διάφορους εκπροσώπους των κρατών. Όχι μόνο δοκιμές αντοχής, αλλά και το μέλλον, προς τα που θα πρέπει να πάμε. Είμαι εναντίον της πυρηνικής ενέργειας και είμαι ε, εναντίον εδώ και δεκαετίες. Αν είχαμε, ε, αν είχαμε ενέργεια, βιομηχανία και τεχνολογία χαμηλού άνθρακα, ε, δεν θα είχαμε ανάγκη την πυρηνική ενέργεια. Ε, και δεν πρέπει να χτίζουμε πυρηνικέ εγκαταστάσει ε, σε σεισμικέ χώρε. Θα πρέπει να μάθουμε το μάθημά μα και από την Ιαπωνία και από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν οπουδήποτε αλλού. Όπω κάνουμε και με άλλε βιομηχανίε. Παραδείγματο χάρη ε, στα σιδηροδρόμου. Υπάρχουν πάντα ατυχήματα. Αλλά κάθε φορά μαθαίνουμε από κάποιο ατύχημα και ε, βάζουμε μέτρα ούτως ώστε το ίδιο ακριβώς ατύχημα να μην ξανασυμβεί. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε όλες τι μορφές παραγωγής ενέργειας πεθαίνει κόσμος, ειδικά στο, στα ανθρακοριχεία α πούμε. Πέθανε κόσμος. Δεν θέλουμε ε, εξαιτίας παλιού αντιδραστήρα του, α, στην Ιαπωνία τελικά να επανέλθουμε ας πούμε ε, στα ανθρακοριχεία και στον, σε μια βιομηχανία που να βασίζεται στον άνθρακα ε, και σε μια ε, τεχνολογία υψηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Λέω κύριο Σλάιτερ. Ε, υπάρχει περίπτωση να κλείσετε κάποιους πυρηνικούς αντιδραστήρες που δεν έχουν ε, προχωρημένα συστήματα ασφάλειας. Επίσης ελπίζω αυτά τα, αυτές οι δοκιμές ε, αντοχής να αφορούν όλη την αλυσίδα. Τη μεταφορά, την, την ε, αποθήκευση ας πούμε, την επεξεργασία του καυσίμου, όλη την αλυσίδα να την τσεκάρετε σε σχέση με τους κινδύνους. Όχι μόνο τους αντιδραστήρες. Έπειτα. Θα πρέπει να κάνουμε μία ανάλυση ε, των καυσίμων. Γιατί το πλουτόνιο, εγώ πιστεύω ότι πάντα ε, εμπεριέχει κινδύνους. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Χθε ε, είπαν ότι αναφέρονται ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σκεφτεί ένα μη πυρηνικό μέλλον. Πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματική σας άποψη και ε, κατά πόσο θα μπορούσαν να, να πιστέψουν οι άνθρωποι κάτι τέτοιο ό,τι αφορά τις δοκιμές αντοχής. Ε, πώς θα γίνονταν αυτές οι δοκιμές ε, για να αποτρέψουμε τις συνέπειες ε, αν ε, παίρνουμε το σχάρι, ε, δούμε τι συνέβη στην Ιαπωνία, το τσουνάμι, ε, τους σεισμούς κτλ. Και αν αποτύχει το, η εγκατάσταση σε αυτή τη δοκιμή, τι θα γίνει. Και λόγω όλων αυτών όπως σκεφτήκατε να υπάρξει ένα μορατόριο για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη μέχρι να έχετε εκπονήσει τις παραμέτρους για τα stress test και να έχουν λάβει χώρα αυτές οι δοκιμές. Ευχαριστώ, Ρώση. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν πολύ ειλικρινεί. Μας είπατε ότι είναι εκτό ελέγχου η κατάσταση. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αποφύγουμε στο μέτρο του δυνατού τις ζημίες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να τροποποιηθεί η ενεργειακή πολιτική της Ένωσης και αν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στη συνθήκη Ευρατόμ. Συγχαρητήρια για την ιδέα σας να ξεκινήσουν αμέσως οι δοκιμές εντοχής, ακόμη και στις ε, φίλες χώρες και ε, να ρωτήσω είναι απαραίτητο από την πλευρά της Επιτροπής να καλέσει τα κράτη-μέλη να ε, μην πάρουν γιαστικές ε, αποφάσεις. Ε, θερμό, θα πρέπει να έχουμε τεχνική υπερογνωμοσύνη για να κατάλαβουμε στην πραγματικότητα ποιοι είναι οι κίνδυνοι και αν αυτοί σχετίζονται μόνο με παλιές πυρηνικές εγκαταστάσεις ή αν σχετίζονται και με τις τελευταίες γενιάς εγκαταστάσεις και αν τελικά θέλετε να κάνετε κάτι για να μειώσετε το κόστο τη ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πρώτον που ήρθατε και δεύτερον το ότι αντιδράσατε τόσο γρήγορα. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι μακροπρόθεσμα θα κάνουμε. Υπάρχει σήμερα μεγάλη πίεση, αλλά σας παρακαλώ, ας κοιτάξουμε μακροπρόθεσμα πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ασφάλεια ε, της ενέργειας ε, και πώς μπορούμε να είμαστε δεσμευτικοί στις αποφάσεις μας. Δεύτερον, θα ήθελα να κοιτάξουμε τα πρότυπα για τις ε, πυρηνικές εγκαταστάσεις Αυτά όλα πρέπει να γίνουν ευρωπαϊκά. Όπως ξέρετε δεν υπάρχουν σύνορα. Όπου και να ανήκει μια πυρηνική μονάδα, οι επιπτώσεις είναι και για τα γειτονικά κράτη και για όλη την Ήπειρο. Δεύτερον, θα ήθελα να ξέρω πραγματικά το πραγματικό κόστος αυτής της ενέργειας και πώς μπορούμε να το υπολογίσουμε. Ματίας Κρότε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά μας δείξατε πως η Επιτροπή μπορεί να είναι αποτελεσματική και να έχει δράση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος συνεχίζει να υπάρχει. Και ο υπολογισμός που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι πότε θα προκύψει κάτι και στην Ευρώπη και αλλού. Δυστυχώς στην Ιαπωνία συνέβη το μοιραίο. Και πολλές φορές αναλύοντας ένα τέτοιο ατύχημα βλέπει κανείς ότι είναι μια λυσίδα συμβάντων που οδηγεί σε αυτήν την κατάσταση, αυτό το ατύχημα. Το ερώτημα που θα κάνουμε σήμερα σε εσά είναι μπορούμε να καταστρέψουμε σήμερα τις υπάρχουσες δομές και την ίδια ώρα να βασιστούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τι μπορούμε να κάνουμε με τα δίκτυα. Τι μπορούμε άμεσα να αλλάξουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα. Είδαμε την ανακοίνωση για την πολιτική προστασία και ως εισηγήτρια θεωρώ ότι θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να τονίσουμε να διευρύνουμε μάλλον ορισμένα κεφάλαια και παραγράφους σε σχέση με το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως ε, να προβλέψουμε για κάποιες προσημειώσεις, ε, κάποια συγκεκριμένα συστήματα πληροφορικής κτλ. Κάτι ακόμη τώρα που θέλω να σας ρωτήσω. Ακούσαμε εδώ για ένα μορατόριουμ. Σήμερα ξέρουμε ότι κατά 30% εξαρτάται από την πυρηνική ενένεια η Ευρώπη και ακόμη και διεθνείς ε, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μας λέει ότι το 2050 θα έχουμε ένα μείγμα μεταξύ ε, αερίων, ενέσιμων πηγών ενέργειας ε, και πυρηνικών. Εσείς ε, τι πιστεύετε σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών. Θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές μέχρι το 2050 χωρίς να έχουμε υποστήριξη από τα πυρηνικά. Ο κύριος Αρσένης. Πολύ σχετική ερώτηση με και αυτή με αυτή της κυρία Τζερντίνη είπατε ότι μπορεί να συμβεί το χειρότερο στην Ιαπωνία και είναι αλήθεια ότι είναι σπάνια τα ατυχήματα σε πυρηνικέ εγκαταστάσει, αλλά όταν συμβαίνουν έχουν πάρα πολύ σοβαρέ διασυνοριακέ συνέπειε και διαρκούν για γενιέ στην ε, προσπάθεια ε, για να μεταβούμε σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050 έχουμε ε, και την πυρηνική ενέργεια μέσα, έχουμε ένα μείγμα και η Κομισιόν έχει κάποια σχέδια, Πώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους μέχρι το 2050 δίχως τη χρήση πυρηνική ενέργεια, ή θα ήταν πρόφημη η Κομισιόν να εκπονήσετε σχέδια κατόπιν του ατυχήματος στην Ιαπωνία. Ευχαριστώ, Κορίν Λεπάζ. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, σας ευχαριστούμε εδώ για την τη δίδρασή σας, την ειλικρινή αντίδρασή σας για το θέμα. Ένα πυρηνικό ατύχημα είναι μια ανθρωπιστική αλλά και οικονομική και χρηματοοικονομική καταστροφή εκτός των μέσων μας ε, φυσικά. Ε, τώρα για το θέμα που τίθεται, ξε, βλέπουμε ότι ό,τι συνέβη στην Επωνία θέλει να ε, ξαναδούμε τους κανόνες κινδύνου, τους τρόπους λειτουργίας μίας εγκατάστασης και να δούμε, και το ανέφερε και ο Πρόεδρος, αν μπορούμε να συνεχίσουμε με μια ρυθμισή όπως αυτή της Ευρατόμ που παρεκκλίνει από το κοινοτικό δίκαιο, θα πρέπει όλα αυτά να τα ξαναδούμε, να βάλουμε μία σειρά και να αλλάξουμε και τρόπους ελέγχου αλλά και κανόνες. Σας ευχαριστώ. Κύριος Ροδρίγες, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας σήμερα και χθε, γιατί σε στιγμές ε, όπως αυτές ε, πρέπει να είμαστε σόφρονες ε, και να μην καταλαμβανόμαστε από πανικό. Σας ευχαριστώ για τις στάσεις σας και για την ταχεία απάντησή σας ε, και επίσης ε, ε, θα ήθελα όλα αυτά να συζητούνται όχι μόνο ε, όταν ψυχ, να μην ξεχαστούν όταν ψυχθούν οι αντιδραστήρες στην Ιαπωνία και να γίνουν αυτές οι δοκιμές εντοχής. Ε, εσείς ε, έχετε πραγματικά σκεφτεί τη δυνατότητα να έχουμε ένα μέλλον χωρίς ατομική ενέργεια στην Ευρώπη και θα είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Κυρία Μπελία. Ευχαριστώ όλοι. Πραγματικά έχουμε σοκαριστεί από τα τραγικά γεγονότα στην Ιαπωνία. Κύριε Επίτροπε, ακούσα ότι προσφύγατε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και συνθήκες για να δικαιολογήσετε μια πολύ μικρή αντίδραση της Κομισιόν. Να σας πω ότι δεν ε, συμφωνώ με την δική σας ανάλυση όταν ε, ε, μιλάτε για την ε, έξοδο από τα πυρηνικά εμείς ε, θεωρούμε ότι θα υπάρχουν συνέπειες. Έχουμε ε, μια γαλλική εγκατάσταση που βρίσκεται ε, σε σεισμική περιοχή και το 2003 με τον καύσωνα είχαμε συνέπειες και φυσικά οι συνέπειες θα είναι για όλες τους Ευρωπαίους. Πιστεύω ότι τα μέτρα ασφαλείας Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε να θέσω την ερώτηση, λέει ο Μιλήτρια. Μα λέτε ότι δεν έχετε την εξουσία, νομίζω την αρμοδιότητα. Νομίζω ότι έχει η Κομισιόν ε, την αρμοδιότητα να τροποποιήσει την νομοθεσία και το ταχύτερο και έχει την αρμοδιότητα να ενισχύσει και να ελοποιήσει αξιολογήσει. Ε, είναι μια παλιά συζήτηση αυτή, αλλά αν το πράξετε αυτό θα σας υποστηρίξουμε. Επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Σόνικ. Δύο σύντομες ε, ερωτήσεις δεν σας προβληματίζει η απουσία του Διεθνούς Οργανισμού ε, Ατομικής Ενέργειας. Δεν ακούσαμε τίποτα από τον οργανισμό για το τύχημα αυτό και δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας ειδικός φόρος για την πυρηνική ενέργεια. Σήμερα τα εργοστάσια λιγνίτη θα πρέπει να αγοράσουν πιστοποιητικά για τις εκπομπές τους. Μήπως θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικοί φόροι, ειδικές εισφορές ε, για τους πυρηνικούς σταθμούς έτσι ώστε να χρηματοδοτούν αντί Πήγες πηγέ ενέργεια. Και η Κριστίνα Γκουτιέρε. Ευχαριστώ. Ε, ε, εδώ ε, πιστεύω ότι λείπουν κάποια λόγια περαιτέρω στήριξης για την Ιαπωνία και βρισκόμαστε ενώπιον μιας καταστροφής που δεν μπορούσε να προβλεφθεί για τον άνθρωπο. Αυτό αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, είχαμε ένα ατύχημα το οποίο κατέστρεψε το σύστημα ψήξη των αντιδραστήρων πολύ συγκεκριμένα. Έτσι νομίζω ότι πρέπει ε, να διαφοροποιήσουμε μεταξύ του τύπου ε, της εγκατάστασης και του ατυχήματος. Το πρόβλημα αυτό ε, ισχύει σε όλο τον ειρηνικό γιατί εκδηλώνονται σεισμοί σε όλο τον ειρηνικό στην Ευρώπη. Όταν χτίζονται τα πυρηνικά εργοστάσια πάντοτε γίνεται μελέτη του εδάφους και να σας πω ότι με πολύ απλό εδώ δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι έχουμε πάρα πολλά πολύπλοκα τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Και μια ερώτηση. Σκεφτήκατε τι κίνδυνο θα δια... Ε... Αν γίνει τέτοιο σεισμός, τι θα γίνει στην Ευρώπη. Ačiū pirmininkė, dėkui komisarė už jūsų tikrai greitą reakciją ir daug sumaišties, daug Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Επίτροπε, για την ταχεία αντίδρασή σας. Πιστεύω ότι αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε την πυρηνική ενέργεια, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε με ασφαλή τρόπο αυτήν την καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε στα σύνορα με την Ρωσία και ξέρετε ότι η Ρωσία στην περιοχή του Καλίνιγκρατ έχει πυρηνικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται να υπογραφεί μια συμφωνία με την Ρωσία και πρόκειται να δοθούν χρήματα στην Ρωσία για την κατασκευή ενός έργου για το οποίο δεν έχει απολύτως καμία συνεργασία με τις γειτονικέ χώρες. Και ήδη η γραμματεία του ΟΣΑ έχει εκφράσει τις ανησυχίες της. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, μιλήσατε για αντίδραση, ταχεία αντίδραση. Συγκεκριμένα, πώς θα τροποποιήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Υπάρχουν πολλές πυρηνικές μονάδες που θα πρέπει να κλείσουν. Σήμερα ξέρουμε ότι οι χειμώνες στην Ευρώπη είναι κρύοι χειμώνες. Είδαμε αγωγούς να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουμε την πυρηνική ενέργεια, να μειώσουμε τις εισαγωγέ μας α, ενέργειας από εξωτερικές χώρες. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτά τα ενεργειακά προβλήματα. Ευχαριστώ. Εδώ και δεκαετίες έχουμε την ε, πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ε, για ποιο λόγο αυτή η καταστροφή στην ε, Ιαπωνία, αυτός ο τρομερός ε, σεισμός ε, είναι κάτι που δεν θα γίνει στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο λόγος που δράτε τώρα κατεπηγόντως σε ό,τι αφορά την προβληματική των Ευρωπαϊκών Πυρηνικών Σταθμών. Εμένα με εκπλήσει η ταχύτητα της αντίδρασης, το επιτακτικός χαρακτήρας, γιατί είδα ότι στην ατζέντα του Συμβουλίου Κορφής την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά δεν γίνεται λόγος για την Λιβύη, εκτός αν έχετε πληροφορίες ε, αλλά εγώ θεωρώ ότι εκεί είναι εκτακ... η κατάσταση είναι έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, γιατί εδώ αντιμετωπίζετε τόσο επιτακτικά αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ, ήσασταν καταπληκτικοί. Και τώρα έχουμε 5-6 λεπτά για τις απαντήσεις. Ο επίγον χαρακτήρας απορρέει από την σημασία της καταστροφής στην Ιαπωνία. Μα τι να σας πω. Είναι κάτι που δεν είναι δυνατόν να το αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο. Σήμερα, πέντε μέρες μετά την καταστροφή, μου προσάπτεται το ότι αντέδρασα επιγόντως. Μα δηλαδή, τι θα μου είχατε πει αν δεν είχαμε κάνει τίποτα αγαπητοί συνάδελφοι. Πραγματικά την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, διότι πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας και η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα αυτά τα συμπεράσματα. Η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ετέθησε ισχύ πριν από ένα χρόνο, δεν πιστεύουμε ότι αύριο θα μπορέσει να ανανεωθεί, να μεταρρυθμιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε τις προσοχές μας σε όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε βάσει παραδείγματος χάρη της συνθήκης γιούρατο. Τι αρμοδιότητες έχουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι εδώ όλες οι σκέψεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η συνθήκη Euratom σήμερα δεν καλύπτει τις αρμοδιότητες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καλύπτει όλα τα θέματα ασφάλειας και πολύ σωστά το φύγουμε το θέμα αυτό. Δεύτερον, το άρθρο 194 και οι αρμοδιότητες για την πολιτική στον τομέα της ενέργειας και αυτό θα πρέπει να το δείξουμε. Και τρίτον, θα πρέπει να πετύχουμε αυτό που δεν πετύχαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά για το θέμα του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Με την στήριξη των κρατών μελών. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι προσπαθώντας να φτάσουμε σε αυτή την ενιαία αγορά θα δημιουργήσουμε και εχθρούς. Γιατί παρόλο που θα μας στηρίξουν οι κυβερνήσεις και τα κράτη-μέλη, θα δημιουργηθούν και αντιπαραθέσεις. Επίσης, οι επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας, που πολλές φορές στηρίζουν και στηρίζονται από τις κυβερνήσεις, δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν να παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Υπάρχουν σήμερα μεγάλες και μικρές πρωτεύουσες δυτικά και ανατολικά που δεν συμφωνούν ακριβώς. Και όσον αφορά την βιομηχανική πολιτική, και όσον αφορά τα μονοπόλια, και όσον αφορά τα καρτέλ, και όσον αφορά τις συμφωνίες για τις τιμές. Δεν θέλουν διαφάνεια, δεν θέλουν ανταγωνισμό και ασφάλεια. Αυτά για μας είναι τα τρία σημεία που βρίσκονται στην καρδιά της δράσης μας. Μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Ενέργειας και θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την περίοδο έτσι ώστε το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά που επιτρέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Με μια διεύρυνση ενδεχομένων των ε, κοινοτικών αρμοδιοτήτων. Μία από αυτές τις αρμοδιότητες που δεν έχουμε και αυτό το αποφάσισαν όντως οι άνδρες και οι γυναίκες πολίτες της Ευρώπης. Το θέμα του μείγματο του ενεργειακού, το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα και στη δική μου περιοχή, στην Βάδεβουρτεμπέργη και εδώ στις Βρυξέλλες, η προσέγγιση όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα είναι διαφορετική. Όντως η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητες για το θέμα αυτό. Εγώ λοιπόν τι μπορώ να κάνω. Να ακούω την Αυστρία με τον Πουρνοκράσκι που δεν έχει πυρηνική ενέργεια και μόνο το 7% της ε, ηλεκτρικής ενέργειας της Αυστρίας προέρχεται από εισαγωγές από γειτονικά κράτη από πυρηνική ενέργεια, ναι. Κατά τα άλλα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διάφορες πηγές πυρηνικής ενέργειας. 7% πολύ καλή αν θέλετε, πολύ καλό μέγεθος. Η Γαλλία όμως έχει 80% που προέρχεται από την πυρηνική ενέργεια. Μεταξύ των δύο λοιπόν εμείς πρέπει να βρούμε μία κοινή θέση. Είναι δύσκολο να φτάσουμε σε ενιαία θέση. Έχουμε την Αρέβα, την ΕΝΤΕΦ, τη Γαλλική Εταιρεία Ελεκτρισμού, χωρίς πυρηνική ενέργεια, τι να σας πω. Επίσης, υπάρχει και η ένταση στην Ιταλία. Εγώ τι να σας πω, δεν έχω δικαίωμα να αποφασίσω για το θέμα αυτό. Όντως δεν υπάρχουν αρμοδιότητες. Όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συνολική ενέργεια που έρχεται από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις 30% σε μέσο όρο. Και βεβαίως για το 2050 έχουμε θέσει κάποιους στόχους. Και για το 2050 ακόμα συζητούμε τους στόχους αυτούς. Όπως προτείνει η Επιτροπή, το 80% των εκπομπών θα πρέπει, μάλλον θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων κατά 80%. Αυτός είναι ο στόχος της Επιτροπής και αυτό θα γίνει μόνο εάν αλλάξει 100% όλη η ενεργειακή πολιτική και μόνο αν μειωθούν κατά 100% οι εκπομπές διοξιδίου. Μηδέν δηλαδή τις 100 εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν έχουμε περιθώριο λοιπόν. Και από σήμερα μέχρι το 2050 θα πρέπει να μην υπάρξει καμία απολύτως ποσοστιαία αύξηση, μόνο μείωση όσον αφορά τις εκπομπές θα πρέπει να υπάρξει. Αλλά βεβαίως ακούτε τι απόφαση ελήφθη στη Γερμανία. Η μεγαλύτερη, αν θέλετε, οικονομία της Ευρώπης. Εάν 7 ή 8 πιο παλιές πυρηνικές, ε, πυρηνικές εγκαταστάσεις σταματήσουν και ξέρετε πολύ καλά ότι η κυρία Μέρκελ δεν είναι ανόητη. Αυτό τι σημαίνει περισσότερη ενέργεια από τον άνθρακα. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Πιστεύω λοιπόν ότι όντως δίπλα στις βραχυπρόθεσμες αυτές δεσμεύσεις και στόχους θα πρέπει να έχουμε και μια μακροπρόθεσμη πολιτική. Ποια είναι η μακροπρόθεσμη αυτή πολιτική όσον αφορά τον ενεργειακό μείγμα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφασίσουν οι υπερογνώμονες αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι μετά από ένα μεγάλο έλεγχο ανθεκτικότητας και δοκιμές αντοχής που θα κάνουμε μετά από αυτά που συνέβησαν στην ε, Ιαπωνία, όλες οι 143 εγκαταστάσεις θα χαρακτηριστούν με θετικό σήμα. Θα κοιτάξουμε αν είναι σεισμογενείς οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται, θα κοιτάξουμε που βρίσκονται σε σχέση με τις πλημμύρες, θα κοιτάξουμε τον εξοπλισμό, θα κοιτάξουμε επίσης και το κόστος. Όλα αυτά είναι τεχνικά, αλλά όχι μόνο. Το καθοριστικό σημείο σε αυτούς τους ελέγχους θα είναι αν το σταμάτημα, το σταμάτημα αυτών των συστημάτων, επίσης των συστημάτων ψήξης, και πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτά που βλέπουμε σήμερα. Γιατί βεβαίως το θέμα της σεισμογένειας της Ιαπωνίας σε σχέση με την Ιαπωνία είναι γνωστό. Αυτό όμως που πρέπει να ελέγξουμε είναι πώς θα επηρεαστεί ή δεν θα επηρεαστεί από άλλους παράγοντες, από παράγοντες δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος παραδείγματος χάρη, το σύστημα ψήξης των ευρωπαϊκών πυρηνικών μονάδων και τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν. Και βεβαίως οι επιθέσεις από αεροσκάφη, τα τσουνάμι ή άλλα φυσικά φαινόμενα, άλλα τεχνικά φαινόμενα. Όλα αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν και να δοκιμαστούν. Πιστεύω και εκεί θα είναι και το κεντρικό σημείο της δράσης μου. Όπως και να βλέπουν τα κράτη-μέλη το ενεργειακό τους μείγμα σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει σήμερα να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα και το πρώτο είναι ότι χρειαζόμαστε σύντομα μία σύγχρονη ευρωπαϊκή υποδομή για την ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτό θα είναι, αν θέλετε, το κεντρικό σημείο αυτού που θα προωθήσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι πραγματικά όσον αφορά το φυσικό αέριο, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, θα συνεχίσουν να υπάρχουν τις επόμενες δεκαετίες. Θα πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν τα πρότυπα, τις δυνατότητες, την ποιότητα και της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και αυτό παντού στον αέριο χώρο και στις πλωτές οδούς και στις θαλάσσιες μεταφορές και στις σιδηροδρομικές μεταφορές, έτσι ώστε και για τους επιβάτες και για τα εμπορεύματα και για τα προϊόντα, για κάθε είδους μεταφορές, τρόφιμα και άλλου είδους εμπορεύματα, οι υποδομές αυτές να αναβαθμιστούν. Το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 20%. Αυτό είναι προϋπόθεση για μας. Και τις επόμενες εβδομάδες θα υποβάλουμε την έκθεσή μας και από εκεί και πέρα βεβαίως πιστεύω ότι λίγοι θα δουν κίτρινη κάρτα ελάχιστη κόκκινη κάρτα και νομίζω ότι το 20% παραμένει η βασική προϋπόθεση. Μέχρι 30%. Και μερικές φορές βλέπω ότι στις μεταφορές είμαστε στο 10%, στις, ε, στην παραγωγή ενέργειας είμαστε στο 30, 33% πολλές φορές αλλά θεωρώ ότι μεταξύ του 20% και του 30% οι επενδύσεις που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικές. Και αν το 2020 έχουμε φτάσει σε πάνω από 30% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 2025, το 2030 θα αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Αυτό είναι το καθοριστικό αν θέλετε. Και με αυτόν τον τρόπο οι εθνικές αρμοδιότητες όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών θα φανεί το πόσο επαληθεύονται. Διότι με αυτόν τον τρόπο οι εθνικές αρμοδιότητες θα μειωθούν. Θα πάνε κάτω από το 60%. Και εκεί θα φανεί πραγματικά ότι χρειάζονται, ότι είναι απαραίτητες σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και στην Ευρώπη, πιστεύω, σιγά σιγά θα αυξηθούν οι νομοθετικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς αυτούς. Όποιος θέλει να προωθήσει και να αναπτύξει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρειάζεται βεβαίως ποδομές, δίκτυα και στόχους κάποια στιγμή να υπάρχει και το οικονομικό αντίτιμο. Το 2011 για μένα είναι καθοριστικό να δημιουργήσουμε έναν χάρτη ευρωπαϊκό που θα συμπεριλαμβάνει και την Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία ε, και την Ορβηγία και την Ελβετία, το Μαρόκο, την Τινησία και άλλες, για μια πανευρωπαϊκή υποδομή, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Καμία άλλη πολιτική δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στον τομέα της ενέργειας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα του ανταγωνισμού. Το δίκαιο του ανταγωνισμού μας θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις παραδείγματος χάρη όσον αφορά την στήριξη που προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Το θέμα βέβαια είναι ότι στον τομέα της ενέργειας χωρίς στήριξη, χωρίς επιδοτήσεις δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και θα πρέπει εδώ να υπάρξουν επενδύσεις τα πρώτα χρόνια που να στηρίζονται, να προβλεφθεί η χρηματοδότησή τους. Αυτό θα το συζητήσω με τον συνάδελφό μου, Αλμούνια. Είναι απαραίτητες αυτές οι στηρίξεις στην αρχή. Και το τραγικό γεγονός που συνέβη στην ε, Ιαπωνία μας δείχνει πραγματικά ότι είτε κανείς είναι υπά είτε είναι κατά της πυρηνικής ενέργειας, αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό σήμερα για όλους μας είναι η ασφάλεια των ε, εγκαταστάσεων που υπάρχουν. Γιατί βεβαίως όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο επικίνδυνη γίνεται η κατάσταση. Και δεν πρέπει να το αναβάλουμε αυτό. Η διεθνής, ο Διεθνής Οργανισμός ε, για την Ατομική Ενέργεια στη Βιέννη, όντως ε, μίλησε πολύ λίγο. Και κατά κάποιο τρόπο παρουσίασε με πολύ ε, σχετικό τρόπο την κατάσταση στην Ιαπωνία. Εγώ την Δευτέρα ζήτησα από το Γενικό Διευθυντή που είναι και η Άπονα εξάλλου. να μας κάνει μία παρουσίαση αυτού του θέματος. Αυτό πάντως που είναι πολύ σημαντικό και θα το επαναλάβω είναι τα πιο αυστηρά πρότυπα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ισχύσουν και να εφαρμοστούν. Και μιλήσατε για το Καλίνιγκραντ, μιλήσατε για τις ε, προσπάθειες της Ρωσίας. Τις παρακολουθούμε. Αλλά είναι σαφές ότι αν ε, αναρωτηθούμε εδώ αν αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα, παράδειγμα, αν παράγεται στη Ρωσία, όπως το φυσικό αέριο, όπως ε, άλλες πρώτες ύλες που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία, μέσω του δικτύου που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να έχουμε και τρόπους πίεσης για αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας. Και βεβαίως στη Λιθουανία οι βαλτικές χώρες, η Πολωνία δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ανταγωνισμό σε όλους τους τομείς, αλλά και στον τομέα της ασφάλειας από το Καλίνιγκρατ, παραδείγματος χάρη. Και αυτό βεβαίως το γνωρίζουμε και σε σχέση με τον σχεδιασμό νέων πυρηνικών αντιδραστήρων στη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητες ε, όσον αφορά τα θέματα της φορολόγησης ε, για αυτούς τους τομείς της ενέργειας. Εξ αυτών θα μπορούσε βεβαίως ε, να προκύψει και μια νέα πηγή χρηματοδότηση, όπως έχει γίνει στη Γερμανία. Εγώ θα έλεγα ότι όντως θα πρέπει να υπάρξει μια ε, φορολόγηση των καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα πρέπει να δούμε αν η πυρηνική ενέργεια βάσει όλων αυτών που θα αποφασιστούν θα αυξήσει το κόστος της, πώς αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που μου κάνατε. Έχω μεγάλη πίεση σήμερα ακόμα μεγαλύτερη μετά την σημερινή συνάντηση. Θα συνεργαστώ όμως με όλους τους ειδικού όλες αυτές τις μέρες και την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για τον καθορισμό αυστηρών προτύπων και την δημιουργία των δοκιμών. Κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. και στηρίζω 100% την ταχεία αντίδρασή σας και εμείς βεβαίως έχουμε εμπειρογνώμονες με μεγάλη χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την θέσπιση ευστηρών προτύπων και για τις δοκιμές αντοχής. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και τα θέματα του κλίματος που και αυτά βεβαίως έχουν σχέση με την ενέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Η κυρία Ρενάτε Ζόμερ. Ηρεμήστε βέβαια πρώτα μετά από αυτήν την πυρηνική ένταση.

Λοιπόν, όποιος δεν θέλει να ακούσει το επόμενο σημείο, μπορείτε να συζητήσετε εκτός της αίθουσας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς θα περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Η Ρενάτε Ζόμερ είναι η συγγήτρια. Θα της δώσω το λόγο. Υπάρχουν τροπολογίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, πάμε στην δεύτερη ανάγνωση. Πρόκειται για τον κανονισμό για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Για τον Ιούλιο έχει προβλεφθεί αυτή η ψηφοφορία και συζήτηση και εμείς θα ψηφίσουμε εδώ τον Απρίλιο στην Επιτροπή, δεύτερη ανάγνωση. Το Συμβούλιο των Υπουργών το Δεκέμβριο πήρε απόφαση, πολιτική συμφωνία. Ήμασταν, θα έλεγα, αρκετά απογοητευμένοι μετά την απόφαση αυτή. Είχαν πάρα πολλές λεπτομέρειες ε, από την πρώτη ανάγνωση, οι οποίες αγνοήθηκαν. Και η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου με την Βελγική Προεδρία μετά από πίεση να βρεθεί συμφωνία υπό Βελγική Προεδρία, εργάστηκε με μεγάλη πίεση χρόνου. Η Ουγγρική προεδρίου πρέπει να σας πω, με βοήθησε να κατανοήσω ορισμένα σημεία. Οι ισχυώδεις εισηγητές ε, συναντήθηκαν με την ε, Ουγγρική Προεδρία συμφωνήθηκε η θέση του Συμβουλίου και θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο καταρχήν θεωρεί ότι το κείμενο αυτού του κανονισμού θα πρέπει να μείνει γενικό έτσι ώστε να καλύπτει πολλά, όσο πιο πολλά ε, σημεία γίνεται που αφορούν τα τρόφιμα. Γιατί θεωρεί ότι όταν παίρνουμε σε πολλές λεπτομέρειες, παραδείγματος χάνει για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα, τα τυριά, ε, γίνονται ειδικέ ε, οι και δεν αφορούν γενικότερα θέματα παραδείγματος χάρη συσκευασίας. Επίσης υπήρξε και κάποιο θέμα ορισμών, δυσκολίες με τους ορισμούς. Επίσης το Συμβούλιο έχει διαφορετική άποψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Όσον αφορά τα προϊόντα που δεν έχουν συγκεκριμένη συσκευασία και ότι αυτά πρέπει να βγουν εκτός του κανονισμού. Παρ' όλα αυτά, η θέση του Συμβουλίου δεν είναι και τόσο κακή σε γενικές γραμμές και όσον αφορά την πρώτη, θέση, την πρώτη ανάγνωση συγγνώμη, και τη θέση του Κοινοβουλίου έχουν ληφθεί υπόψη αρκετά σημαντικά Στη μία πήγαν 170 τρυπολογίες και όντως βλέπουμε ότι έτσι όπως έχει συνήθως η κατάσταση αυτός ο αριθμός είναι αρκετά ε, Τώρα, το δικό μου σχέδιο. Σας είπα καταρχήν ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να καθορίσει την έννοια του, της συσκευασίας, της εξωτερικής συσκευασίας. Πολλές φορές υπάρχουν ε, προϊόντα που έχουν, ε, αν θέλετε, διάφορες επιφάνειες συσκευασίας, διάφορες όψεις, όπως τα ποτά, παραδείγματος χάρη. Το θέμα λοιπόν της ποια είναι η εξωτερική όψη επιφάνεια, τι φαίνεται, παραδείγματος χάρη, μέσα στο μαγαζί από τον καταναλωτή και εδώ αυτό είναι πολύ δύσκολο να οριστεί. Ποια είναι η όψη. Ε, το θέμα είναι πού βρίσκεται ο καταναλωτής τελικά, από ποια πλευρά βλέπει ε, ένα πακέτο. Το θέμα τώρα της, του ευανάγνωστου χαρακτήρα, του πόσο εύκολο είναι να κατανοήσει κανείς ή να διαβάσει αυτήν την συσκευασία. Και εδώ υπήρχαν διάφοροι περιορισμοί. Η Επιτροπή ζήτησε να καθοριστούν ε, και άλλες προδιαγραφές. Υπάρχει ο ορισμός της Επιτροπής για την αναγνωσιμότητα. Αλλά πραγματικά τα κριτήρια αυτά είναι αρκετά περιοριστικά. Το σημείο 7, το άρθρο 7, η παραπλανητική ενημέρωση. Εδώ υπήρξε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση και πιστεύω ότι εδώ, ακριβώς επειδή πολλές φορές υπάρχουν ελλειπείς πληροφορίες, λείπει παραδείγματο χάρη ένα πολύ σημαντικό συστατικό. Εδώ, παραδείγματο χάρη όσον αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά ή σε ζάχαρη ή σε θερμίδες, ο καταναλωτής πολλές φορές, άμα λείπουν κάποια στοιχεία, μπορεί να θεωρήσει ότι επειδή υπάρχει λίγη ζάχαρη, είναι χαμηλός και ο ε, αριθμός των θερμίδων. Εδώ λοιπόν αυτό το θεωρούμε παραπλανητική ενημέρωση. Το Συμβούλιο δεν θέλει όμως παρόλα αυτά να μπει ε, μέσα σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις λέγοντας παραδείγματος χάρη τι είναι ε, καινοτομία, τι είναι απομίμηση, τι είναι τι είναι οι απομιμήσεις και αυτό βεβαίως ε, ε, εδώ το είχαμε ορίσει εμείς την πρώτη μας ανάγνωση. Επίσης, η προσθετική προστιθέμενες ουσίες και οι απαγορευμένες ουσίες. Σε σχέση με την ποσότητα βεβαίως στην οποία περιέχονται. Ε, ο, το μέγεθος ε, όσον αφορά τα γράμματα που χρησιμοποιούνται, όλα αυτά είναι καθορισμένα. Εδώ Επίσης μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για τα κατεψυγμένα προϊόντα η ημερομηνία κατάψυξης και αυτό θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο. Και εδώ επιμείναμε πολύ για το μέγεθος των γραμμάτων που χρησιμοποιούνται. Μπορεί να είναι τεχνικό το θέμα, αλλά εμείς θέλουμε όλα αυτά να ληφθούν υπόψη, γιατί είναι και αυτό το τμήμα του, της αναγνωσιμότητας για τα υνοπνευματόδη. Εμείς είχαμε προτείνει να φύγουν ε, τα προϊόντα αυτά, τα, τα, η κατηγορία των Alcopops είναι όλα αυτά τα προϊόντα που είναι μείγματα μεταξύ υνοπνευματοδών και μη. Άλκοποψ αυτά θα πρέπει κανονικά να συμπεριλαμβάνουν και μείγματα με μπύρα και μείγματα με κρασί. Τελικά όμως είδαμε ότι η Επιτροπή έχει ε, ορίσει τελείως διαφορετικά τα προϊόντα αυτά και εδώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Επιτροπή. Άρα λοιπόν τα αλκοπόψ δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε, την, ε, σε αυτό το κείμενο. Ή επιπλέον ε, αξίες. Εδώ συμφωνεί μαζί μας το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να υπάρχει σήμανση σε γραμμάρια, σε λίτρα και όχι σε μονάδες που δεν τις κατανοεί παραδείγματος χάρη ο καταναλωτής. Να μιλάμε σε θερμίδες και όχι σε τζάουλ. Αυτό είναι κάτι που πάντα δημιουργεί σύγχυση. Επιπλέον όμως θα πρέπει να υπάρχει περιεκτικότητα σε θερμίδες, σε πρώτη θέση και κατόπιν να υπάρχει σε μία παρένθεση ή περιεκτικότητα σε τζάουλ. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι θερμίδες και στην εμφανή όψη, αν θέλετε, ε, των προϊόντων και αυτό να είναι υποχρεωτικό και με αρκετά μεγάλα γράμματα. Αυτό υπήρχε στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και υπάρχει και στον κόντεξ αλιμετάριους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα πρέπει να αποκλειστούν. Επίσης τα προϊόντα τα βιοτεχνικά, αυτά βεβαίως αποκλείονται. Και όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, τα εποχιακά προϊόντα, και αυτά αποκλείονται. Το θέμα της προέλευσης, εγώ είμαι υπέρ να αποφύγουμε εδώ κάποιες πολύ προστατευτικές ε, τάσεις κάποιων κρατών που αν θέλετε έχουν πάρα πολύ περιοριστικές ε, ρυθμίσεις. Η Ιταλία παραδείγματο χάρη που ζητάει να υπάρχει η μνήα, η αναφορά της προέλευσης, της εθνικής προέλευσης. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, έτσι κι αλλιώς ε, θα πρέπει εδώ να γίνει μια μελέτη αντικτύπου, να δούμε αν αυτό επηρεάζει συγκεκριμένα τις επιλογές. Η Επιτροπή θεωρεί βεβαίως ότι μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και πολλά άλλα στοιχεία, το Συμβούλιο Υπουργών, όσον αφορά την προέλευση, κάτι που είχε ισχύσει παραδείγματος χάρη για το κρέας, και είχε ήδη αποφασιστεί. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις έχουν ε, ήδη αποφασιστεί ανατομέα. Επιπλέον τώρα ρυθμίσεις για το κρέας, για προϊόντα κρέατος, χωρίς ε, μελέτες αντικρύπου. Αυτό το έχουμε απορρίψει και νομίζω ότι το Συμβούλιο εδώ ζητάει ε, αξιολόγηση. Τελειώνοντας, το Συμβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει σήμανση στην, στην ε, μπροστινή όψη όλων αυτών των συσκευασιών για θέματα ενέργειας σε θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Ελπίζω επιτέλους το Συμβούλιο να συμφωνήσει μαζί μας σε αυτό που το ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και επιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σόμερ για την παρουσίαση αυτών των τροπολογιών, για τη δεύτερη ανάγνωστη. Από ό,τι φαίνεται σε πολλά σημεία υπάρχει σύγκληση. Αυτόν δηλαδή που στηρίξαμε στην πρώτη ανάγνωση και την κοινή θέση του Συμβουλίου παραμένουν κάποια θέματα εκκρεμή. Έχω ένα κατάλογο ομιλητών. Κένις Βίλμοτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Ζόμερ για την πρόσκληση να συναντηθώ με την Ουγγρική Προεδρία. Ήταν πολύ χρήσιμο, την ευχαριστώ. Ε, έχω πολλά να πω για τη θέση του Συμβουλίου. Ε, πολλά είναι καλά, αλλά θέλω να επικεντρωθώ σε τρία βασικά θέματα. Γιατί η θέση του Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα ήταν ξεκάθαρη. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα που θα είχα προβλήματα. Τα τρία βασικά μου προβλήματα που θέλω να αναφέρω είναι τα εξή. Καταρχά, είναι εμπρόστια όψη. Η θέση του Κοινοβουλίου ήταν ξεκάθαρη ότι θα πρέπει να έχουμε τα, τα πέντε βασικά θρεπτικά στατικά μπροστά. Συμφωνώ, κυρία Σόμερ, ότι οι εξηγήσει του Συμβουλίου που δεν τα βάζουν προς την επρόστια όψη, ας πούμε, είναι γελία. Θέλουμε λοιπόν τα πέντε βασικά στατικά μπροστά, ε, ας πούμε λίπη ε, και κορεσμένα λίπη, α, καλωρί, ζάχαρη κτλ. Ούτω ώστε ο κόσμος να βλέπει αμέσως τους πέντε, τα πέντε βασικά θρεπτικά στατικά ε, στα τρόφιμα. Επίσης, ε, δεύτερο θέμα είναι η χώρα προέλευσης. Ε, το Συμβούλιο συμφώνησε να υπάρχει επισήμαση σε όλα τα ψάρια και τα κρέατα. Ε, η θέση του Κοινοβουλίου επίσης ήταν ξεκάθαρη. Είμαι στεναχωρημένη όμως που δεν πετύχαμε την επισήμαση της χώρας ε, προέλευσης σε μεταποιημένα ψάρια και κρέας. Ε, αφού το έχουμε στα φρέσκα, γιατί όχι και στα μεταποιημένα, δεν το καταλαβαίνω το επιχείρημα είναι, ας πούμε, αν αγοράσω ε, σάντουιτς κοτόπουλου στο Ενωμένο Βασίλειο και λέει παράγεται στο Ενωμένο Βασίλειο, το, το σάντουιτς όμως, αλλά το ε, κοτόπουλο ε, παράγεται στην Ταϊλάνδη, ας πούμε. Έχουμε θέματα και ευημερία των ζώων, ας πούμε, α, για κρέατα που παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε κανόνες, αλλά όχι στο εξωτερικό. Ε, υπάρχει και το θέμα του τρόπου μεταφορά. Και επίση οι καταναλωτέ θέλουν να ξέρουν από πού προέρχεται, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και το μετοποιημένο κρέα. Επομένω, θέση του Κοινοβούλου ήταν σαφή και γι' αυτό. Ε, επίσης, ε, τα λιπαρά τρανς. Τα λιπαρά τρανς. Εθελοντική λέει αναγραφή το Συμβούλιο, δεν μου αρέσει αυτό. Ξέρουμε ότι οδηγούν σε προβλήματα γονιμότη, ε, γονιμότητας, Αλτσχάιμερ, σε καρδιακά προβλήματα κτλ. Αν έχετε δύο τρόφιμα που είναι ίδια από διαφορετικούς παραγωγούς, ο ένας εθελοντικά βάζει το περιεχόμενο σε λιπαρά τρανς και ο άλλος δεν λέει τίποτα, παρόλα αυτά περιέχει όμως το ε, το τρόφιμο αυτό λιπαρά τρανς, ο, ο καταναλωτής πιστεύει ότι αυτός που δεν λέει τίποτα, ας πούμε, είναι πιο, ε, έχει πιο υγιεινό, α, πιο υγιεινή τροφή, ας πούμε, αγοράζει αυτό, αλλά αυτό είναι παραπλανητικό, δεν είναι σωστό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Εντάξει, να βάλουμε μία απαγόρευση, αλλά το... δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Μέχρι να φτάσουμε στην απαγόρευση όμως θα πρέπει να αναγράφονται και τα λοιπά τρανς. Ε, υπάρχουν πολλά άλλα θέματα ε, επομένως θα πω... Αυτά μάλλον ήταν τα τρία βασικά θέματα. Ε, δεν, θα είχα πολλά ακόμα να πω, αλλά θέλω να μιλήσουν και άλλοι. Το βασικό είναι να δίνονται πληροφορίες μέσω αυτής της επισήμανσης στους καταναλωτές. Είναι κάτι που το λέω συνέχεια. Αν θέλουμε να δίνουμε πληροφορίες στους καταναλωτές, ούτως ώστε να κάνουν υγιεινές περιπτώσει, επιλογές, εφόσον το θέλουν, για αυτούς και για τις οικογένειές τους χρειαζόμαστε ξεκάθαρη επισήμανση. Επομένω, σκεφτείτε το Σκεφτείτε την εμπρόστια όψη των τροφίμων, τα λιπαρά τρανς και ελπίζω να μετακινηθεί προς τη δική μας θέση το Συμβούλιο ε, σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ, Γκλένης. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επανέρχομαι στην πρώτη ανάγνωση. όπου εκεί παίξαμε πόλεμο χαρακομμάτων. Το Συμβούλιο έκανε μία προσπάθεια μετά, ε, δέχτηκε διάφορες συμβιβασμούς και μάλιστα βρήκε και συμβιβασμούς που δεν μπορούσαμε εμείς να βρούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για αυτή την προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, οι φιλελεύθεροι δεν είναι ε, σύμφωνοι με όλα όσα πρότεινε το Συμβούλιο. Αλλά, εν πάση η θέση του Συμβούλιου βοηθάει. Συμφωνώ με δύο από τα τρία στοιχεία. Κυρία Χέλμουτ. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λοιπόν συνέκλειναν. Καταρχά συμφωνώ με την κυρία Βίλμουτ σε ό,τι αφορά τα λιπαρά τραν. Είναι πολύ σημαντικά, πολύ ανθυγινά για να τα ξεχάσουμε στην ε, επισήμανση. Επομένως θα υπάρξει τροπολογία για αυτό. Συμφωνώ με την κυρία Ζω, Σόμερ και την κυρία Βίλμουτ σε ό,τι αφορά την οπίστια όψη της συσκευασία. Δεν συμφωνώ με το Συμβούλιο που λέει ότι σε ορισμένες περιπτώσει δεν είναι σημαντική η όψη αυτή. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στην ε, θέση του Κοινοβουλίου της πρώτης ανάγνωσης για τους πέντε, τα πέντε βασικά συστατικά στην εμπρόστια όψη και όχι μόνο την ε, θερμιδική αξία, όπως είπε η συγγήτρια προηγουμένως. Και πάω τώρα στην χώρα προέλευσης. Δεν θα σε εκπλήξει βέβαια ότι δεν πάω τόσο μακριά όσο η κυρία Βίλμουτ. Οι φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι υπάρχει εσωτερική αγορά. Στο, παρελθόν υπήρχαν επιτακτικοί λόγοι να αναφέρουμε στο βόλιο κρέας την χώρα προέλευση. Υπήρχαν λόγοι. Τώρα όμως, εφόσον έχουμε εσωτερική αγορά, για ποιο λόγο να έχουμε αυτή τη διάταξη και για άλλα είδη κρέατος. Μπορεί να γίνει θελοντικά, εντάξει. Αλλά εμείς πιστεύουμε στην αγορά. Αν ο εμπορο στην αγορά πιστεύει ότι μπορεί να πείσει περισσότερο το καταναλωτή, αναφέροντα ότι το κρέα του είναι από, το, από τη Γαλλία, από το Βέλγιο ή το Ηνωμένο Βασίλειο, α το κάνει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εντάξει, επειδή είχαμε και, έχουμε και μεγάλη πλειοψηφία στη δεύτερη ανάγνωση, ε, αποφασίσαμε ως φιλελεύθεροι να δεχτούμε ενδεχομένως τη θέση, να κουνηθούμε, εν να αλλάξουμε και να, δεχτούμε, να κινηθούμε προς τη θέση του Συμβουλίου. Για την ε, ημερήσια συστηνόμενη δόση τώρα. Δεν υπάρχει υποστήριξη στο Κοινοβούλιο για την αναφορά αυτή τη συνιστόμενη ημερήσια δόση ή πρόσληψη. Αν πούμε στον καταναλωτή ότι υπάρχουν τρία γραμμάρια αλατιού, το τάδε προϊόν, τι σημαίνει αυτό. Αν δεν ξέρει, α πούμε, πόσο, πόσα γραμμάρια αλατιού μπορεί να φας την ημέρα. Είχαμε μία θέση στην πρώτη ανάγνωση. Είχαμε ένα σύστημα που ήταν κατανοητό για από τον καταναλωτή. Αλλά πώς θα μπορέσει ο καταναλωτής να γνωρίζει μόνο τον αριθμό των γραμμαρίων, να καταλάβει αν είναι υγιεινό, αν είναι καλό ας πούμε αυτό το φαγητό ή όχι. Το σύστημα που λέει πόσο πρέπει να καταναλώνουμε την ημέρα, χοντρικά ας πούμε, αυτό είναι μια καλή ένδειξη, χρήσιμη για τον καταναλωτή. θα υποβάλω και σχετική τροπολογία και ελπίζω να μπορέσω να πείσω και τους συναδέλφους των άλλων ομάδων και ελπίζω να τους πείσω να το ξανασκεφτούν και να μετακινηθούν. Τέλος πάντων, τώρα το προϊόν που προέκυψε χάρη στο Συμβούλιο είναι πιο ευανάγνωστο, πιο εύληπτο από αυτό της πρώτης ανάγνωσης. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την παρουσίαση. Μπορώ να συμφωνήσω με τα σχόλια των ομιλητών ε, για την προστινή όψη του πακέτου. Όσοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα τραφήμα, ξέρουμε ότι εύκολα ε, κάποιο αναγνωρίζει την προστινή όψη του πακέτου. Έτσι λοιπόν πρέπει οι πληροφορίε να βρίσκονται σε αυτή την προστινή όψη και πρέπει να μείνουμε στην αρχική μα θέση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χώρα προέλευση. Ήδη υπάρχει αυτό για το βόλιο κρέα, αλλά για λόγους διαφορετικούς από τη σημερινή συζήτηση. Και επομένω υπάρχει ενδιαφέρον μεταξύ των καταναλωτών να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων κρέατος και σε σχέση με τις ανησυχίες που ακούστηκαν για το μετοποιημένα τρόφιμα, ίσως υπάρχει μια συνέπεια αν κάπου έχουμε την προέλευση, ενώ σε άλλα σε άλλα προϊόντα όχι. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο θέμα σε ό,τι αφορά τα αποψυγμένα προϊόντα. Ε, ίσως να το αναφερθεί σε αυτό και η συγγήτρια, ίσως δηλαδή χρειάζεται τα προϊόντα να φέρουν ε, αυτή την ε, ετικέτα ε, που είναι αποψηγμένα. Νομίζω ότι οι ορισμένα κρατημπέλη υπάρχουν, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα και υπάρχει σύγχυση γιατί υπάρχει αυτή η ετικέτα και αν είναι απαραίτητη για να ενημερώνεται ορθά ο καταναλωτή. Ελπίζω να έχουμε μια πιο εύκολη δεύτερη ανάγνωση, αλλά ήθελα να ξεκαθαρίσω αυτά τα συγκεκριμένα σημεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το σκιώδη εισηγητή που είναι στον μου. Παίρνω το λόγο εκ του. Νομίζω ότι η δεύτερη ανάγνωση, τουλάχιστον από τη σκοπιά του Κοινοβουλίου, θα είναι κάπως πιο εύκολη. Νομίζω θα μπορέσουμε πιο εύκολα να καταλήξουμε στα κυρία σημεία. Βέβαια, πότε δεν ξέρει και κανείς, αλλά ας είμαστε θετικοί. Α είμαστε αισιόδοξοι, γιατί εμείς τα τρία κυρία σημεία που έχουμε εμεί ω πράσινοι είναι τα κυρία σημεία που αναφέραν και άλλοι συνάδελφοι, η κυρία Βίλμουτ, με χάρη, ε, τώρα για τους πρασίνους ε, το κύριο θέμα είναι η υποχρεωτική αναγραφή ε, των στοιχείων στην προστιμίωση του πακέτου. Δεύτερον, η υποχρεωτική σήμανση των λιπαρών τρανς. Αν δείτε τι σημαίνει την νομοθεσία, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υποχρεωτική αναγραφή των λιπαρών τρανς και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κάτι θέση. Τρίτον, χώρα προέλευση ίσως χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό με του φιλελευθέρου, αλλά τελικά νομίζω ότι εμείς συμφωνήσαμε στο Κοινοβουλίο ότι η χώρα προέλευση είναι ζωτική σημασία για τον οίκο αυτό. Και μιλάμε και για τα μεταποιημένα τρόφιμα, παραδείγματο χάρη, αν έχουμε τρία τρεις χώρες, δηλαδή γέννηση του ζώου, ε, εκτροφή και σφαγή, πρέπει να αναγράφονται και αν ε, εμείς ε, τώρα στο Κοινοβούλιο μένουμε σε ορισμένα θέματα, πρέπει να διατηρήσουμε την ισχυρή θέση μας στη δεύτερη ανάγνωση και να έχουμε ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Μάριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να κάνω τρία σχόλια επί ορισμένων ε, τροπολογιών που παρουσίασε η κυρία Ζόμερ. Για την τροπολογία 15. Για την 70. αναφέρονται στις ε, διατροφικές ε, τιμές για 100 γραμμάρια, έτσι όπως καταγράφεται εδώ, προϊόντος, παραδείγματος χάρη για 100 γραμμάρια. Έτσι, όπως ε, καταγράφεται εδώ, θεωρώ ότι εμείς μπερδεύουμε τον καταναλωτή. Γιατί όταν πρόκειται, παραδείγματος χάρη, για ένα προϊόν 100 γραμμαρίων, εντάξει. Αν όμως το πακέτο συμπεριλαμβάνει και μερίδες, τότε δεν ε, νομίζω ότι ε, βοηθούμε τον καταναλωτή. τόσο χάρη στα κράκερ. Ε, μέσα σε ένα πακέτο κράκερ μπορεί να υπάρχουν ε, μεμονωμένε μερίδε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα και οι πληροφορίε, οι διατροφικέ, πρέπει να αναφέρονται οι πληροφορίε, διατροφικέ για τη μερίδα. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει αυτό να ισχύει για κάθε συσκευασία. Δεύτερον, Θέλω να ρωτήσω την μου πώς μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει τροπολογία 19, όπου λέει ότι τα προϊόντα μη προσυσκευασμένα που, προκα... που πολλούνται προσωπικά στον ε, ε, καταναλωτή και μπορεί να, παρουσια... να δημιουργήσουν δυσανεξία ή αλλεργίες πρέπει να ε, δίνονται γι' αυτό προφορικές πληροφορίες. Ε, δεν ε, καταλαβαίνω ακριβώς τι σημαίνει αυτή η τροπολογία. Μήπως θα έπρεπε να βάλουμε ουσιαστικά κάτι διαφορετικό εδώ. Τώρα, τροπολογία 23 αποκλείεται από τα προσκευασμένα προϊόντα, τα συσκευασμένα στο σημείο 20. Αυτό μπορεί να ισχύει για τις ε, συσκευασίες όταν είναι παρόν ο καταναλωτής, αλλά όχι όταν ε, ε, δεν παρευρίσκεται ο αγοραστής. Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει παρόλα αυτά να περιλαμβάνουν πληροφορίες στην ετικέτα. Διαφορετικά δεν ε, θα σεβόμαστε το στόχο που έχουμε θέσει, δηλαδή να προστατεύσουμε το καταναλωτή σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την εισηγήτρια θα είμαι σύντομη σε ό,τι αφορά την δήλωση των διατροφικών στοιχείων, οι πληροφορίες για τις θερμίδες και για τα ε, θρεπτικά στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν στην προστινή όψη ανά 100 γραμμάρια και 100 μιλιλίτρια. Δεν είμαι πεπισμένη από τη θέση ε, της εισηγήτριας εδώ ε, θα πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι τι αγοράζουν. Δεν είναι θέση τη βιβλίο Τώρα, για τα λιπαρά τρανς, ε, στη δική μας πρόταση, στην πρώτη ανάγνωση είχαμε κάνει, ε, είχαμε υποβάλει μια πρόταση που πρέπει να τη διατηρήσουμε για τη χώρα προέλευσης η κοινή θέση του Συμβουλίου δεν ε, είναι απόλυτα απορριπταία, πρόκειται για ένα πρώτο βήμα. Νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο αυτόν τον κανόνα. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση Ηνωμένων συναδέλφων, δηλαδή να έχουμε ε, υποχρεωτική αναφορά ε, της προέλευσης για τα μεταπημένα προϊόντα για την Ασπαρτάμι έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Εμείς προτείνουμε για τα προϊόντα που περιέχουν ασπαρτάμι να αναφέρεται ότι περιέχουν ασπαρτάμι και σε παρένθεση πηγή φαινενολενίνης και αναρωτιέμαι αν μήπως θα έπρεπε και μία σύσταση εδώ για τις εγκύους για τα πρόσθετες μορφές έκρησης ε, ε, θα πρέπει η Επιτροπή να παρουσιάσει μια έκθεση για τη θέση εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι πολύ μακρά αυτή η παράγραφος. Θα καταθέσω τροπολογία για τη σύγκριση και να σα πω ότι κατά τα λοιπά συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε εδώ η κυρία Βελιμούτα Ευχαριστώ κυρία Λέπας. Θα πρέπει να συνηθίσω ότι είναι συντονιστής. <laughs> Κύριε Ρώση, ευχαριστώ. Η επιτέθηκε στην Ιταλία γιατί θέλει πάρα πολλές συνδείξεις προέλευσης για να ε, προστατεύσει τις τυπικές παραγωγές της. Έτσι, λοιπόν, ε, έχουμε χώρες όπως η Ιταλία που έχουν τέτοια τυπικά προϊόντα, σαλάμια, τυριά, γλυκά, ε, αν ε, επιτρέψετε κάτι τέτοιο όπως είχαμε το φανάρι, αν ξαναμπεί δηλαδή τώρα κάτι που βγει από την πόρτα από το παράθυρο ή ε, τη δυνατότητα να έχουμε διάφορες συνδείξεις ε, και να έχουμε παραδείγματος χάρη ένδειξη και αναμερίδες. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι κανένας δεν τρώει 100 γραμμάρια ε, ή 80 ε, γραμμάρια λαδιού, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το βάλουμε για τα 100 γραμμάρια για να ε, φοβήσουμε τον καναλωτή. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ε, δηλαδή, αν ε, τώρα σε ένα ρούχο μπροστά του του τυπώσουμε από τι αποτελείται, κανείς δεν θα το αγοράσει, γιατί είναι το ίδιο. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά εμείς ε, θα καταστρέψουμε αυτόν τον τρόπο την συσκευασία του προϊόντος. Αν άνθρωπος, ε, κάποιος αγοραστής ενδιαφέρεται για το τι τρώει, θα γυρίσει το προϊόν και θα διαβάσει τις ε, πληροφορίες στην ετικέτα από την πίσω πλευρά. Και έτσι θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία 23 και στην Λιρογόνα και αυτές οι τροπολογίες είναι παράξενες. Εγώ συμφωνώ όμως, είπε ο συνάδελφος Σπυρίλο, γιατί φαίνεται ότι ε, μοιάζουν με κάτι που πρότεινε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και τελικά πρόκειται να ευνοήσει το μεγάλο σούπερ μάρκετ που τι κάνουν, αγοράζουν το προϊόν και στη συνέχεια ε, αυτοί το συσκευάζουν και το βάζουν στα ράφια προς Και αυτά τα σούπερ μάρκετ ε, δηλαδή δεν χρειαζόταν καν να βάλουν την ετικέτα με αυτροπολογία. Πολύ ιδιάζουσα η επιλογή σα εδώ, αν θέλετε, να βοηθήσετε τον καταναλωτή και το ίδιο και για τις αλλεργικές ουσίες και πάντε. Ε, πάντοτε εδώ θα έπρεπε, παραδείγματο χάρη, οι άνθρωποι που πουλούν αυτά τα προϊόντα, όταν πάει ε, ο αγοραστή εκεί, να του πούν ε, αν προκαλεί αλλεργία το προϊόν. Κοιτάξτε, και το McDonald's ακόμη έχει και τον κατάλογο με τις αλλεργογόνες ουσίες τα προϊόντα του. Όμως για την εισηγήτρια, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ μπορούν να συσκευάζουν αγοράζουν και να πολλούν χωρί ετικέτα και χωρί καμία ένδειξη για τι αλλεργιογόνες ουσίες. Ε, όμως ε, μας ζητήσατε ε, άλλα πράγματα όπως η σήμαση προέλευσης. Τώρα κοιτάξτε την ένδειξη του ύψου των ουσιών του περιεχομένου ε, μάλλον της γραμματοσυράς σα το αποφασίσει η Κομισιόν. Δηλαδή τελικά θα έχουμε τεράστιες ετικέτες για τις ε, ενδείξεις ε, προέλευσης του είπε. Εμείς είμαστε υπέρ, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε να πούμε στον καταναλωτή τι τρώει, από πού ε, προέρχεται, για τα 100 γραμμάρια τοποθετήθηκα, είναι ε, υπερολικό, οι θερμίδες πρέπει να δίνονται αναμερίδα για τις ελεγγονωσίες, το είπα. Μεραμένει το θέμα που έθιξε ένας άλλος συνάδελφος, το οποίο συμφωνώ εμείς. Ε, ε, εδώ αν είναι μεικτό το προϊόν, δεν μπορούμε να αναφέρουμε την ημερομηνία κατάψυξη του προϊόντο. Σα σκεφτείτε μία ψαρόσουπα, παραδείγματο χάρη, μεικτά λαχανικά που έχουν 10, 15, 20 προϊόντα διαφορετικά στην ίδια συσκευασία. Πώ θα υπάρχει ένα κατάλογο 20 διαφορετικών ημερομηνιών κατάψυξη για κάθε προϊόν, γιατί διαφορετικά καταψύχεται το κάθε προϊόν και παράγεται σε διαφορετικό χρόνο. Παραδείγματο χάρη το ψάρια ή διαφορετικά φρούτα, διαφορετικά λαχανικά. Είναι αδύνατον. Ε, δηλαδή, σίγουρα η ημερομηνία που θα αναγράφει την ημερομηνία λήξη. Δεν μπορούμε να μιλάμε εδώ για ε, την αναγραφή 20 ημερομηνών κατάψυξη στη συσκευασία. Λυπάμαι που το κείμενο αυτό ε, ίσως ε, αποτελεί επιδείνωση σε σχέση με το κείμενο που πέρασε στην πρώτη ανάγνωση. Εμείς θα παρουσιάσουμε μια σειρά τροπολογιών ε, για να βελτιώσουμε το κείμενο. Ελπίζουμε να εγκριθούν διαφορετικά. Ε, σίγουρα θα καταψηφίσουμε. Merci. Ε. Ευχαριστώ κύριε Ρώση. Φρεντερικ Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ διαφωνώ με την αυστηρότητα του συναδέλφου Ρώση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σόμερ, η οποία δεν τα πέτυχε όλα βέβαια, αλλά τουλάχιστον κατάφερε τις φιλόδοξες προτάσεις μας εδώ στην πρώτη ανάγνωση. Πολλές φορές δεν ήμασταν και πολύ λογικοί, δεν είχαμε μεγάλη συνοχή, αλλά ήμασταν τουλάχιστον φιλόδοξοι και η κοινή θέση, η συμβαστική αυτή θέση, σε γενικές γραμμές είναι καλή. Αν και αρκετά γενική, όπως είπε και η συγγήτρια. Κάτι με το οποίο συμφωνώ είναι η αναφορά του κράτους προέλευσης. Εγώ στηρίζω την πρόταση του Συμβουλίου. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει η αναφορά και για το γάλα και για το κρέας, τα κλερικά και κάποια άλλα προϊόντα που δεν αποτελούνται από πολλά διαφορετικά συστατικά. Νομίζω ότι ο καταναλωτής θέλει σήμερα να γνωρίζει ε, από πού προέρχονται τα προϊόντα που αγοράζει, αλλά είναι και πολύ σημαντικό για τις περιοχές που έχουν παραγωγές, ειδικέ παραγωγές και αν εγώ πάω να ψωνίσω σαν ε, Ευρωπαίος καταναλωτής, ε, θέλω να γνωρίζω αν μια ντομάτα που αγοράζω προέρχεται από το βορρά, γενικά λέω τώρα το βορρά, ή μια ωραία ιταλική ντομάτα με ωραία γεύση. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά μας αφορούν η πράσινη βίβλο στην οποία ήμουν και εισηγητής εξάλλου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία. Είδα ότι επίσης για τα λιπαρά τρανς δεν συμφωνεί η Επιτροπή, ούτε από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο, τουλάχιστον τα φυσικά λιπαρά τρανς που υπάρχουν σε κάποια γαλακτοκομικά προϊόντα και σε κάποια προϊόντα κρέατος και στα λιπαρά τρανς που δεν είναι φυσικής προέλευσης. Τουλάχιστον εδώ να υπάρξει μία διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών και στην τροπολογία 144 υπήρχε αυτή η ε, αναφορά. Η Επιτροπή προτείνει έξι υποχρεωτικές ε, αναγραφές. Εμείς έχουμε μια λίστα οκτώ. Ας επιμείνουμε σε αυτές. Θα ήθελα να πω στην εισηγήτρια και τελειώνω ότι, όπως είπε η εισηγήτρια, διαφωνεί να υπάρχει η αναγραφή για ένα προϊόν το οποίο λείπει, παραδείγματος χάρη. Προϊόντα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μία αλλεργία, είναι αλγογόνα προϊόντα. Κατάλαβα καλά τι είπατε, θα ήθελα μία διευκρίνηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Άζα Όσλουν έχει το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί που είπαν ότι θα πρέπει οι αναφορές αυτές να γίνονται στην προστινή όψη του πακέτου της συσκευασία έχουν δίκιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διατροφική αξία, τα συστατικά, την χώρα προέλευσης. Η κυβέρνηση της Σουηδίας θεωρεί ότι, και δεν είναι η μόνη βεβαίως, ένας ε, καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ξέρει από πού προέρχεται το κρέας που αγοράζει. Αυτό είναι προφανές. Και ο καθένας θα πρέπει να μπορεί να διαλέξει το κρέας του και να ξέρει από πού προέρχονται και τα ε, ζώα από τα οποία παράγεται το κρέας, αλλά και τα προϊόντα κρέατος και τουλάχιστον τα βασικά συστατικά θέλουμε να ξέρουμε από πού προέρχονται σε μεταποιημένα προϊόντα. Υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης έτσι ώστε αυτά τα οποία αναφέρονται στις συσκευασίες να είναι όντως ορθά. Αυτή είναι μια ερώτηση. Δεύτερον, όσον αφορά τα λιπαρά τρανς, σήμερα η κυβέρνηση της Σουηδίας έχει απαγορεύσει αυτές τις κατηγορίες ε, προϊόντων. Και καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθούν δυσκολίες αν δεν υπάρχει ομοιόμορφη νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαγόρευση λοιπόν για τα λιπαρά τρανς, αυτή είναι η δική μας θέση. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό δεν περάσει, να υπάρχει αναφορά με σαφέστατο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει ο καταναλωτής εγώ πιστεύω και επιμένω ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται ορθά για το τι θέλει να αγοράσει. Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι στην έκθεση Ζόμερ, πέρα από τις πληροφορίες που δίνουμε στους καταναλωτές, θα πρέπει να αναφερθούμε και στην ποιότητα των τροφίμων. Πιστεύω ότι οι δύο κανονικοί, θα οι νέο κανονισμοί συγγνώμη, θα πρέπει σήμερα να εναρμονιστούν. Εγώ ήμουν σκιώδης εισηγητής για το θέμα αυτό της ποιότητας και υπάρχουν σαφώς επικαλύψεις. Βλέπω πολλές επικαλύψεις και πολλές δυσκολίες, πολλές αντιφάσεις. Παραδείγματο χάρη δεν υπάρχει ενα, εναρμόνιση όσον αφορά την ποιότητα και όλων των υπόλοιπων αναφορών που προβλέπει ε, η κυρία Ζόμερ στην έκθεσή της. Επίσης, ε, ιδιαίτερα με ενδιαφέρουν τα μεταποιημένα προϊόντα στην Επιτροπή Γεωργίας. Υπάρχει, η υπάρχει σαφής πλειοψηφία όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα, τρόφιμα, για τα οποία θέλουμε να υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, η χώρα προέλευσης, ο τόπος προέλευσης. Και γι' αυτό η Επιτροπή Γεωργίας είναι υπέρ σε μεγάλη πλειοψηφία. Θέλω επίσης να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα των υνοπνευματοδών ε, ποτών. Εγώ είχα πολλές συζητήσεις με την ε, βασίλισσα, αν θέλετε, ε, του κρασιού και των προϊόντων αυτών, την κυρία Λούλινγκ. Γιατί, παραδείγματος χάρη, δεν βάζουμε τις θερμίδες, την περιεκτικότητα του κρασιού σε θερμίδες. Και αυτό θα μπορούσαμε να το βάζουμε σε ένα μπουκάλι κρασί. Και για άλλα είναι ο πνευματόδη. Δεν ξέρω, κρίμα δεν είναι. Υπάρχει ένα λόμπι εινοπαραγωγών που πραγματικά απαγορεύει κάτι τέτοιο. Εμένα μου αρέσει το κρασί, πίνω κρασί. Αλλά γιατί δεν επιτρέπουμε μια τέτοια ρύθμιση. Επίσης θεωρώ ότι η προθεσμία των τεσσάρων ετών είναι πολύ μεγάλη πρέπει πραγματικά να επανέλθουμε στο σύστημα του κόκκινου, κίτρινου και πράσινου σηματοδότη. Στην Ουγγαρία, στην εποχή του κομμουνισμού, υπήρχε ένα παρά, παρόμοιο ε, σύστημα και πρέπει να σας πω ότι ο καταναλωτής ήταν υπέρ, γιατί είχε μεγάλη πληροφόρηση για τα τρόφιμα, για το θέμα του σηματοδότη θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να επανέλθουμε σε 8 χρόνια. Σε 3 χρόνια θα πρέπει το Συμβούλιο να έχει επανέλθει στο θέμα αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχει επιθυμία από την κοινή γνώμη για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροτ Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάτι σε δύο διαφορετικά σημεία αυτής της έκθεσης. Αυτά που είχαν στηριχθεί στην πρώτη ανάγνωση πρόκειται για θέματα τα οποία θα ήθελα με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να πω ότι ένα προϊόν θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές θα πρέπει να φαίνονται τα συστατικά, τα βασιστάτικα, συστατικά, όπως είπε η κυρία Βέσλου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί εδώ να συμβιβαστούμε. Δεν θα αλλάξουμε τη θέση μας και στην κοινή θέση με το Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικό αυτό που υπάρχει και το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν θέλουμε μόνο για τα προϊόντα χοιρινού κρέατος αλλά και τα πουλερικά να ξέρουμε την προέλευση. Θέλουμε μια γαρίδα να ξέρουμε αν είναι από το Βόρειο Ατλαντικό, από τη Μεσόγειο ή από την από Ανατολή. Γιατί πραγματικά δεν είναι θέμα παραπλάνησης, είναι θέμα νομοθεσίας. Το θέμα λοιπόν του άρθρου 25, εδώ σε αυτή την κοινή θέση, που μιλάει για τη χώρα προέλευσης, είναι μη ικανοποιητικό, θα το πω έτσι. Επίσης, το θέμα της κοινή θέσης όσον αφορά τις ποσότητες, τα 100 γραμμάρια και στο άρθρο 100 βλέπω ότι λέγεται ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να αναγραφεί και η αξία αναμερίδα. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί ή δεν μπορεί. Εγώ είμαι πολλά χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο και ποτέ δεν είδα μέχρι τώρα στη δεύτερη ανάγνωση μια έκθεση να μην αντικατοπτρίζει την πρώτη ανάγνωση. Κυρία Ζόμερ, πολύ ειλικρινά θέλω να σας πω και δεν με ενδιαφέρει τι θεωρείτε εσείς. Εάν κοιτάξει κανείς την πρώτη και τη δεύτερη ανάγνωση, ο καθένας μπορεί να πει τι νομίζει και τι θέλει, αλλά δεν έχει πλέον σημασία. Εσείς είστε δεσμευμένοι από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Πάει, πέταξε το πουλί. Δεν είναι πλέον δική σας η έκθεση. Είναι έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είστε συγγήτρια, αλλά πλέον το θέμα εναπόκειται στην Ολομέλεια. Και αυτήν την εντολή έχετε. Όσο δίκιο και να έχετε, σας παρακαλώ πολύ, πρέπει να υλοποιήσετε την αποστολή σας, να εκπληρώσετε την αποστολή σας βάσει αυτών που ισχύουν. Δεν είναι λοιπόν η δεύτερη ανάγνωση πραγματικά σε ε, ομοφωνία με την πρώτη ανάγνωση. Και το θεωρώ σκανδαλώδες. Όποια και να είναι η δική σας άποψη, δεν μπορείτε εδώ να δέχεστε αυτή την κατάσταση. Αλλιώς υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Μπορείτε να βρείτε συμβιβασμούς. Εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλά τίποτα άλλο δεν μπορείτε να κάνετε. Αλλιώς θα υπάρξει επίσημη διαμαρτυρία. Merci. Euh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρουτ Μπέρεντ. Η κυρία Γκαρντίνη. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια σημεία από τα οποία παρουσίασα τροπολίες διάφορα πράγματα υπόθηκαν ε, με τα οποία συμφωνώ. Πιστεύω ότι η ετικετοθεσία αναμερίδα είναι σημαντικό, επισήμαση αναμερίδα. Παραδείγματος χάρη μπισκότα. Αν εγώ το πρωί, ε, το πρωινό μου είναι ένας καφές και τρία μπισκότα, θέλω να ξέρω κάθε μπισκότο πόσα καλωρί μου δίνει, πόσε θερμίδε μου δίνει. Δεν μπορώ να μου λέτε εσεί, α πούμε, τα 100 έχουν τόσο και να αρχίσω να κάνω διαιρέσει, α πούμε, για να βρω πόσο έχει το μπισκότο, πόσε θερμίδε. Θέλω να ξέρω πόσε θερμίδε τρώω με κάθε μπισκότο. Εντάξει. Ο καναλωτή θέλει την ε, ενημέρωση αυτή ανά μερίδα. Οπότε, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την αναγνωσιμότητα. Καλό θα ήταν να αφήσουμε σε ένα κανονισμό, ο οποίος μπορεί να αλλάξει αν αλλάξουν οι συνθήκες, αυτό το θέμα, αντί εμείς να μπούμε σε λεπτομέρειες. Γιατί η αναγνωσιμότητα, όπως ξέρετε, έχει να κάνει όχι μόνο με το μέγεθος των χαρακτήρων των γραμμάτων, αλλά και με πολλά άλλα πράγματα. Εγώ έχω παρουσιάσει τροπολογίες που μου φαίνονται πιο αποδεκτές. Επίσης, αυτό που είχαμε εγκρίνει εξαφανίστηκε, αν δεν απατώμε. Το θέμα των ιδιωτικών ε, ετικετών. Αυτό εξαφανίστηκε. Νομίζω είναι θέμα διαφάνειας απέναντι στον καταναλωτή. Αν η επιχείρηση, ας πούμε, διανομής αλλάζει προμηθευτή, λογικό είναι ο καταναλωτής να ενημερωθεί. Θα έπρεπε. Ε, ενώ όμως αυτό ε, κρύβεται μέσα στο σήμα, ας πούμε, του διανομέα. Δεν είναι σωστό αυτό. Επίσης, για τα αλλεργιογόνα. Όλη αυτή η συζήτηση με έχει μπερδέψει. Θέλω να μάθω πώς λειτουργεί το όλο πράγμα. Γιατί είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο το ποσοστό δηλαδή των πολιτών που παρουσιάζουν αλλεργίε. Και ξέρετε τι, πόσο δραματικές είναι οι συνέπειες. Μερικές φορές καταλήγουν, οδηγούν και στο θάνατο οι αλλεργίε. Επομένω, είναι πολύ λεπτό το θέμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να εντοπίζονται τα αλλεργιογόνα. Αν υπάρχουν, αναφέρονται λοιπόν. Επίσης, πιστεύω ότι τα ε, προϊόντα που συσκευάζονται επί τόπου, εκεί όπου πολλούνται, δεν θα πρέπει να μας οδηγούν σε αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν είναι λόγος για αθέμητο ανταγωνισμό. Συνολικά, πρέπει να έχουμε μια στάση πιο θετική, πιο ενεργητική. Ε, απέναντι στη δυνατότητα του καταναλωτή να διαχειριστεί την πληροφορία όλα αυτά, πληροφορίες μπροστά, πίσω στο πακέτο, όλα αυτά είναι υπερβολικό, γιατί δείχνουν πραγματικά μια δυσπιστία απέναντι στην ικανότητα του καταναλωτή να καταλάβει τι τρέχει. Και απ' την άλλη, το να ξαναβάλουμε το μικρό παραθυράκι, όπως υπόθηκε, το, την ετικετοθεσία ε, σαν το ε, σήμα της κυκλοφορίας. Αυτό είναι σαν το φανάριμα της κυκλοφορίας. Αυτό είναι προβληματικό. Ε, μην ξεχνάμε τα προβλήματα που έχουν πολλοί έφηβοι, ας πούμε, με την τροφή. Αν βάλουμε, ας πούμε, μπροστά στο, στην όψη του πακέτου, ε, ξέρω εγώ, ένα φανάρι με κόκκινο, ας πούμε. Δημιουργούμε προβληματική σχέση. Ε, τα καρότα είναι πολύ υγιεινά, έχουν πολλέ θετικέ ουσίε. Όταν τρώει κανεί μόνο καρότα, α πούμε, είναι κακό. Χρειάζεται μια ε, κουλτούρα, α πούμε, ε, διατροφή για να είμαστε υγιεί. Πριν από δύο εβδομάδε έγινε μια διάσκεψη ενό σημαντικού ε, πανεπιστημιακού που έλεγε ότι θέλω να ξέρω το θερμιδικό περιεχόμενο ενός τροφίμου. Δεν πρέπει εμείς να μπούμε σε λεπτομέρειες με τρόπο γελίο που οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, θα μας μισήσουν. Θα μας μισήσουν. Αν καθίσουμε εκεί πέρα σε ένα σύννεφο θεωρητικό, ας πούμε. Δεν πρέπει να οδηγήσουμε σε ένα μίσος ε, προς την Ευρώπη τους πολίτες. Μια Ευρώπη, θα πρέπει αντίθετα να προωθήσουμε μια Ευρώπη και να αγαπήσουμε μια Ευρώπη που είναι κοντά στους πολίτες, ε, μια Ευρώπη, α πούμε, να προωθήσουμε την Ευρώπη των διαφορετικών πολιτισμών κτλ. Να μην τα φοβόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Ο επόμενο ομιλητή. Κύριο Σνέλχαρτ, ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Νομίζω ότι έχει διαρκέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν συμβιβαστική λύση και αν κάποια θεωρούνται ότι αγνοήθηκαν παρόλα αυτά. Έτσι γίνεται πάντα σε κάποιους συμβιβασμούς και σε όλους τους συμβιβασμούς εξάλλου. Στην πρώτη ανάγνωση δεν μπορούμε να διατηρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση όλο το περιεχόμενο της πρώτης ανάγνωσης. Τι να σας πω, αυτό το θέμα πάντως το συζητάμε εδώ και χρόνια. Και είναι πολύ αρνητικό αν, όπως παραδείγματο χάρη απορρίφθηκαν κάποια σημεία ε, από την πρώτη ανάγνωση στη δεύτερη, εμείς να προσπαθούμε να τα επαναφέρουμε. Ε, κάτι που ουσιαστικά δεν θα βοηθήσει να υπάρχει μεγάλη υποψηφία. Η σήμανση στον μπροστινό ή στο πίσω τμήμα του πακέτου της συσκευασίας. Κοιτάξτε, και εδώ έγινε προσπάθεια συμβιβασμού. Το σημαντικό είναι να ενημερωθεί ο καταναλωτής, έτσι δεν είναι. Και η προσωπική μου άποψη είναι, όταν πηγαίνω να αγοράσω, κοιτάω ουσιαστικά ποια είναι η ανάγκη μου για κάθε χρόνο και σε τι ποσότητα ανταποκρίνεται αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να πιέσουμε και να ενισχύσουμε τις προτάσεις μας. Πρέπει να δείξουμε ευελιξία. Ρυθμίζονται τα περισσότερα θέματα. Ο ευανάγνωστος χαρακτήρας αυτών των ε, πληροφοριών, ναι, το μέγεθος των γραμμάτων, ναι. Και Βεβαίως δεν συμφωνούμε σε όλα εδώ, αλλά το θέμα της προέλευσης σε κάθε περίπτωση μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Ίσως το παρατραβάμε. Η αναφορά στη χώρα προέλευσης για κρέατα, παραδείγματος χάρη, δικαιολογείται. Αλλά, τι να σας πω, να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση και οπωσδήποτε πρέπει να ξέρουμε τη χώρα προέλευσης όλων των προϊόντων. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι στην Ευρώπη τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας, ότι δεν προκαλούν προβλήματα για τη δημόσια υγεία. Τώρα μην είμαστε και υπερβολικοί. Γιατί αν θέλουμε, παραδείγματο χάρη, να πούμε ναι, αυτό είναι από τον τόπο μας, αγοράστε το, να το κάνουμε. Αλλά να μην υπάρχει υποχρέωση αναγραφής δεσμευτική. Και α είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε η πληθώρα πληροφοριών στις ετικέτες να μην δημιουργήσει σε περισσότερη σύγχυση έτσι ώστε οι σημαντικές πληροφορίες να χαθούν μέσα στις πολλές πληροφορίες. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι η υποχρεωτική αναγραφή του χώρου, της χώρας προέλευσης είναι λίγο υπερβολική έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κορίν. Λέω ο κύριος Ουτζίας. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάνουμε καλή δουλειά στην Ολομέλεια. Αφαιρέθηκαν πολλά σημεία από την αρχική θέση. Η, η έκανε καλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να το βελτιώσουμε περισσότερο το κείμενο. Θα τη ζητούσα λοιπόν να δείξει ανοιχτό πνεύμα ε, σε προτάσεις βελτίωσης. Γιατί πρέπει να συνεργαστούμε. Όχι να συγκρουστούμε όπως κάναμε επί κάποιων τροπολογιών της πρώτης ανάγνωσης. Υπήρξαν ε, προτάσεις βελτιωτικές από πλευράς του Συμβουλίου, να τις λάβουμε υπόψη μας. Και θέλω να ξαναπροτείνω το εξής. Να επαναλάβω ουσιαστικά μια κριτική που είχα διατυπώσει την πρώτη ανάγνωση, που αφορούσε την επισήμανση της χώρας προέλευσης. Τη χώρα λοιπόν προέλευσης. το να αναφέρουμε την τάδε χώρα, αυτό είναι πολύ γενικό λόγο. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση όπου μιλάμε για... Συχνά μιλάμε, ας πούμε, για την πολιτιστική, οικονομική αξιοποίηση, ας πούμε, διαφόρων περιοχών. Έτσι. Χρήσιμο δεν θα ήταν, λοιπόν, να εξειδικεύσουμε και τις επισημάσεις μας, να προτάξουμε αυτή την προστιθέμενη αξία που έχουν πολλά προϊόντα συχνά είναι εδαφικά σήματα. Ε, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ποιότητα, σημαίνει προσθέμενη αξία για την υγεία. Μου άρεσε λοιπόν η τροπολογία του Συμβουλίου προς αυτήν την κατεύθυνση, η παριθμόν 82. Κυρία Βίλμοτ και κύριε Ρώση, δείτε την. Λέμε ότι θα αφήσουμε στη χώρα προέλευσης ή στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να εισαγάγουν διατάξεις που να αφορούν την υποχρεωτική ένδειξη της χώρας προέλευσης ή του τόπου από τον οποίο προέρχονται τα τρόφιμα. Μόνο όταν υπάρχει σύνδεσμος αποδεδειγμένος με την ποιότητα του, μεταξύ της ποιότητας του τροφίμου και της α, χώρας δεν μπορούν όλες οι χώρες Φερρυπίν να βάλουν ας πούμε ένα σήμα περιφερειακό. Όταν υπάρχει ποιότητα, όταν υπάρχει προστιθέμενη αξία, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει στο σήμα, να φαίνεται με το σήμα. Μέσα σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας θα ήταν ένα ερώτημα ε, στην εισηγήτρια. Αν θέλετε να μου απαντάτε. Για ποιο λόγο προτείνετε τη διαγραφή της τροπολογίας 82 του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Και περιμένω την απάντηση βέβαια. Ευχαριστώ. Κυρία Χιμπνερ. Ευχαριστώ. Ή Χίμπνερ καλύτερα. Ευχαριστώ. Ακόμα μια φορά σήμερα κοιτάμε ένα θέμα όπου είχαμε συνένεση στην πρώτη ανάγνωση. Το Συμβούλιο έκανε τροπολογίες με διαφορετική διατύπωση που νομίζω ότι διαστρεβλώνει την, το κείμενο που υιοθετήθηκε στην πρώτη ανάγνωση. Η πληροφορία για τους καταναλωτές θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη, τελεία και τίμια. Ε, και πλήρης. Δεν είναι θέμα μόνο μεγέθους. Είναι και θέμα αντίθεσης γραμμάτων και χρώματος της συσκευασία. Εξαρτάται από το χρώμα αυτό, εάν τα γράμματα τελικά είναι ευανάγνωστα ή όχι. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες προς τους καταναλωτές είναι όσο να τον πιο προσπελάσιμες. Δεύτερον, δεν συμφωνώ με τους συναδέλφους που μειώνουν τη σημασία της χώρας προέλευσης. Πολλά προϊόντα προέρχονται από χώρες όπου οι διαδικασίες παραγωγής είναι τέτοιες που δεν θα άρεσαν στους καταναλωτές. Παραδείγματο χάρη ε, μεταποιημένα τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα. Πολλοί, μπορεί να μην θέλουν να υπάρχει αυτή η πληροφορία, ας πούμε. Έπειτα, χρειαζόμαστε ένα συμβιβασμό ε, για την θερμιδική αξία. Μπορούμε να έχουμε ε, την αξία ανά 100 γραμμάρια ή 100 ml ή αναμερίδα, την τιμή μάλλον των θερμίδων. Εξαρτάται πώς παρουσιάζεται. Τα 100 γραμμάρια είναι καλή, καλό μέγεθος αναφοράς για ορισμένα προϊόντα. Αλλά για άλλα προϊόντα που έχουν συγκεκριμένες μερίδες ή μεγέθη, ας πούμε, όπως ακούσαμε από την κυρία Γκαρντίνη, τα μπισκότα, ας πούμε, δεν έχει νόημα να πει θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Θα βάλεις τώρα έναν ηλικιωμένο να κάνει διαιρέσεις για να βρει πόσα, ε, πόσες θερμίδες ε, έχει το συγκεκριμένο μπισκότο, ας πούμε θα πρέπει να δίνουμε ξεκάθαρες και τίμιες πληροφορίε στους καταναλωτέ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ. Να μιλήσω για τι αλλεργίε. Δεν μιλήσαμε πολύ, ε, πολύ για τις αλλεργίες. Ε, σαν πολιτικός θα πρέπει να σταθώ σε ατομικές περιπτώσεις, όμως θα να πω το εξή. Στην πρώτη ανάγνωση είχα υποβάλει μια τροπολογία. Την 24, αν θυμάμαι καλά. Και την δυνατότητα να γράψουμε μπορεί να περιλαμβάνει ίχνη αλλεργιογόνων ουσιών. Φοβόμουν ότι μια πολύ αυστηρή νομοθεσία θα μπορούσε να παραβλέψει α, σημαντικές πληροφορίες. Εγώ, ας πούμε, είμαι ε, αλλεργικός στα φουντούκια. Στα καρύδια, συγγνώμη. Ε, εγώ, ας πούμε, επειδή δεν έχω μεγάλη αλλεργία, ε, μπορώ να φάω κάτι που έχει ίχνη α, καρυδιών. αλλά αν ήταν πιο σοβαρή η αλλεργία μου, δεν θα μπορούσα ούτε αυτό να ανεχτώ. Εγώ δεν λέω ότι, ότι στο, σε ένα συγκεκριμένο ας πούμε, προϊόν έχουν μπει επίτηδες ε, καρύδια, αλλά θα μπορούσαν να είχαν μπει ε, χωρίς να το θέλουμε ίχνη, να υπάρχουν ίχνη χωρίς να το θέλουμε. Ένα άλλο επίμαχο θέμα. Έχει πλάκα πάντα να μιλάς για επίμαχα θέματα για το ενόπνευμα. Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό να βάλουμε το περιεχόμενο σε ενόπνευμα. Και όχι σε θερμίδες. Μπορεί κάποιος να διαλέξει, ας πούμε, να πάρει ένα προϊόν με ενόπνευμα γιατί πιστεύει ότι έχει λίγες θερμίδες. Θα πρέπει να το δούμε χωριστά, στα πλαίσια μιας παρέκκλησης στο θέμα του ενόπνευματος. Ένα άλλο θέμα πολύ επίμαχο. Σε διάφορες αποφάσεις, το ΔΕΚ είπε ότι οι εθνικές προδιαγραφές με τις ε, με την ονομασία προέλευσης βάζουν εμπόδια, ας πούμε, στο εμπόριο. Ε, ξέρω, ας πούμε, ότι το καλύτερο κρέας είναι το σουηδικό, ενώ το χειρότερο είναι το δανέζικο, το, το βουλγάρικο, ας πούμε. Η ονομασία προέλευσης θα πρέπει να γίνεται θελοντικά. Δεν χρειάζεται να νομοθετήσουμε ε, επί του θέματος αν ε, οι επιχειρήσει ε, το θέλουν να το χρησιμοποιήσουν αυτό σε επιχείρημα για να ανταγωνιστούν η μία την άλλη, οκ. Για τα ψάρια. Δεν θέλουμε να είναι ε, θολή η ένδειξη, ας πούμε, της ονομασίας προέλευσης. Ας πούμε, από τον Ανατολικό Ατλαντικό. Τι σημαίνει αυτό. Αν θέλουμε να βάλουμε υποχρέωση για τα ψάρια, τουλάχιστον ε, να δίνει ξεκάθαρη πληροφορία που προέρχεται το συγκεκριμένο ψάρι. Όχι γενικολογίες. Και τελευταίο και σημαντικό. Η κυρία Γκαρντίνη, προηγουμένως, είπε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα της απλούστευσης. Ε, και μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος δεν είναι ανόητος. Ε, δεν σημαίνει ότι αν αν μπει ας πούμε κάτι στην οπίστια όψη, δεν σημαίνει ότι ο, ο, ο καταναλωτής δεν θα βρει την πληροφορία. Θα τη βρει την πληροφορία, γιατί δεν είναι χαζός. Φυσικά ο καθένας είναι και υπεύθυνο για τη σωστή χρήση αυτών των πληροφοριών. Ε, δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να μπουν πάντως στην εμπρόστια όψη. Α, ο καταναλωτής μπορεί να βρει πληροφορίες και μπρος και πίσω. Ευχαριστώ. Λέει κυρία Βενίνο. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε ευθύνη και για τις επόμενες γενιές ε, και φυσικά για τη δική μας αλλά και για τις επόμενες γενιές ο καλύτερο, το καλύτερο μέσο να ε, παράσχουμε εμπιστοσύνη στον καταναλωτή για τα προϊόντα είναι να είμαστε διαφανείς και να αναφέρουμε τις πληροφορίες. Και δεν μιλάμε για θέμη του ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών. Νομίζω ότι είναι καθήκον για τον καταναλωτή που αγοράζει. Πρέπει να γνωρίζει τι αγοράζει και από πού προέρχεται. Είναι σημαντικό ακριβώς για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Γιατί όταν γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι αγοράζουμε από τη Δανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία κτλ. Δεν ξέρουμε και επιλέγουμε. Και αυτό εκπαιδευόμαστε. Και κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι μια περιοχή από τα Δυτικά και συχνά συζητώ με του αλείς του Δυτικού Ατλαντικού ε, και συναντώ και αλληλείς ε, μη επαγγελματίες αλλά και όσους έχουν και μεγάλα σκάφη και μου λένε ότι ε, και οι ίδιοι κάνουν και μπορούν να ε, αναφέρουν από πού προέρχεται το ψάρι. Εδώ συμφωνώ με τον εντελώ συναδέλφο ότι είναι σημαντική προέλευση και για τι περιφέρειε. Υπάρχουν συγκεκριμένε περιφέρειε ε, που είναι σημαντικό να γράφεται η περιφέρεια για την ποιότητα των προϊόντα και όταν μιλάμε για ταφική συνοχή, ε, για δημιουργία θέσεων εργασία στι περιφερειέ μα και για καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, ε, θα πρέπει να μπορούμε να προσδώσουμε αξία σε μια περιφέρεια και να βλέπουμε για τα φρούτα και τα λαχανικά αν ε, παραδείγματο χάρη σεβόμαστε και όλα όσα θέλουμε να κάνουμε για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Αγοράζουμε τώρα στα φύλλα από τη χιλή το Δεκέμβριο. Τι να σα πω, ναι, μπορεί να το διαλέξει ο καταναλωτή, αλλά την περασμένη παραδείγματο χάρη Κυριακή ε, ήθελα εγώ να αγοράσω γλυκάνισο. Πινόκιο. Πινόκιο και ήρθε από την Κίνα. Δεν ήθελα λοιπόν ε, να, αγοράσω ένα προϊόν από τόσο μακριά γιατί θεωρούσα ότι δεν ήταν υπεύθυνο από περιβαλλοντική σκοπιά. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να αναγράφεται αυτό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να στείλει πάρα πολύ ισχυρό σύμπα, ισχυρή θέση το Κοινοβούλιο σε αυτή τη δεύτερη ανάγνωση. Έτσι λοιπόν ε, ε, πρέπει να, είναι επιτακτικό να ζητήσουμε και την απαγόρευση των τεχνητών λιπαρότρας και για τις αλλεργεγόνες ουσίες. Ε, βλέπουμε ότι αυξάνονται οι αλλεργίες στα παιδιά και στους εφήβους. Πρέπει να υπάρχει απαραίτητη σήμανση. Κατόπιν για το θέμα τη μερίδα. Νομίζω ότι μπορούμε να αναφέρουμε την ποσότητα των λιπαρών, των σακάρων, ε, του αλατιού ε, και όταν έχουμε συγκεκριμένε μερίδε, όπω τα μπισκότα να αναφέρουμε τι θερμίδε και για τι ε, μερίδε. Παραδείγματο χάρη μπορούμε να αναφέρουμε πόσε θερμίδε έχουν τα τέσσερα μπισκότα. Πρέπει όμω να είναι όλα αυτά διαφανή και απλά. Γιατί εδώ μιλάμε και για εκπαίδευση. Και ε, φυσικά ξέρετε ότι η εκπαίδευση καλύπτει πολλές πολιτικές. Ευχαριστώ κύριε Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, ο Γιώ είπε ότι οι απόψει σε αυτήν εδώ την Επιτροπή είναι μακριά από την ομοφωνία. Θα ήθελα παρόλα αυτά εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί όντως αυτή τη δεύτερη ανάγνωση βλέπουμε διαφορές μεταξύ του κειμένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτού του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι είναι δύσκολη η δουλειά της εισηγήτριας και έκανε πολλά για να φτάσει σε αυτό το κείμενο. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Συζητούμε εδώ πολλές διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις και ακούσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε την αξία, τη θερμιδική αξία αναμερίδα, ανακομμάτι. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ αυτού. Θα ήταν καλό για όλους να είχε κανείς την αξία για λιγότερο από 100 γραμμάρια 100 ml και να μπορεί ο καταναλωτής να διαπιστώσει πόσες θερμίδες, πόση ενέργεια έχει μια μικρότερη ποσότητα, μια μικρή μερίδα ή ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Και μια άλλη παρατήρηση θα ήθελα να κάνω όσον αφορά τις ενδείξεις για την προέλευση ενός προϊόντος. Σαφώς και υπάρχουν ε, χώρες που με πολύ εύκολο τρόπο μπορούν να βάλουν την ε, ένδειξη για τη χώρα προέλευσης για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Πολύ δύσκολα όμως θα το πετύχουμε αυτό όταν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα είτε για προϊόντα που περιέχουν πολλά διαφορετικά συστατικά, πολλά διαφορετικά είδη. Αυτό σαφώς θα σημάνει πολύ μεγάλο κόστος για αυτόν που παράγει το τελικό προϊόν. Θέλουμε βεβαίως να υπάρχει προστασία του καταναλωτή, θέλουμε όμως μια απλοποιημένη διαδικασία η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πλήξει και δεν θα περιπλέξει τη δουλειά του παραγωγού. Η Λίντα. Ευχαριστώ. Δεν ε, πρόκειται να πάρω το λόγο, αλλά θέλω να αφαιρθώ σε κάποια σημεία που ακούστηκαν αναφερθήκατε στην ε, σήμαση της χώρας προέλευσης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η σημερινή νομοθεσία για τη χώρα προέλευσης μπορεί να οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή, γιατί το κρέας μπορεί, παραδείγματο χάρη, να φέρει την ε, ετικέτα της χώρας της τελευταίες μεταποίησεις ε, ή συσκευασία. Μπορείτε, παραδείγματο χάρη, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Όταν ρώτησα την ε, Κομισιόν μου είπαν ε, οι Βρετανικές Αρχές αυτό το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου είπαν όχι είναι Βρετανική Νομοθεσία που έχει κάνει ε, αυτό το λάθος και υπάρχει λοιπόν στο νόμο μία ένα κενό που πρέπει να το κλείσει η νομοθεσία. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε την παραπλάνηση των καταναλωτών. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για τα ψάρια. Οπότε καταλαβαίνω, ήδη ούτως ή άλλως φέρουν ετικέτα τα ψάρια ήθελα να επανέλθω σε είπε ο Ντάγμαρ και να ζητήσω από την ε, κυρία Ζόμερ να δει την ε, πρώτη ανάγνωση. Εκεί έχουμε ε, συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υποχρεωτική σήμαση της προέλευσης και για τα πέντε θρεπτικά στοιχεία και ε, υποχρεωτική σήμανση για τα λιπαρά τρανς. Αυτές τις τελειθέσεις μας ε, νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθούν στη δεύτερη ανάγνωση σε ό,τι αφορά τώρα τις μερίδες εναντί των 100 γραμμαρίων. Σε πολλά προϊόντα και τα δύο υπάρχουν και είναι πολύ απλό. Νομίζω ότι μπορούμε να συμβαστούμε με το Συμβούλιο για να έχουμε και τα δύο. Ο λόγος για τον οποίο δεν αρκεί ε, η μερίδα είναι γιατί μπορεί παραδείγματο χάρη να πει ο, ο ε, ότι αυτό είναι για τέσσερα άτομα, ενώ κάποιοι αυτή την ποσότητα μπορεί να τη φάνε δύο άτομα. Έτσι λοιπόν ε, ξέρω παραδείγματο χάρη ότι έχουμε 60 μερίδες ε, να αναγράφονται σε πακέτα δημητριακών και αν ρωτήσετε μια οικογένεια φυσικά δεν θα φάνε 60 φορές από αυτό το πακέτο γιατί θέλει φυσικά ο κατασκευαστής να ελκυστοποιήσει το μέγεθος της μερίδας για το αλκοόλ. Καθόμουν στο τρένο της προάλλες και έπινα εγώ χυμό πορτοκάλι και ο άντρας μου μπήρα. Εγώ είχα όλες τις θερμίδες στο κουτάκι του χυμού για τις θερμίδες, τα σάχαρα ενώ στην πύρα του τίποτα δεν αναγραφόταν. Και ξέρετε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κατανάλωση αλκοόλου στην Ευρώπη. Οι νέοι πίνουν πάρα πολύ, πολλά ένα πνευματόδη. Έχουμε πρόβλημα παχυσαρκία. Πρέπει, παίρνουμε το σχάρι, να ενημερώσουμε του ανθρώπου ότι αν πίνουν τέσσερα ποτήρια κρασί είναι το ίδιο με το να φάνε ένα γεύμα. Και δεν θα καταστρέψουμε τη χαρά του να πιει κάποιο κρασί, απλώ θα συνειδητοποιεί τι ακριβώ καταναλώνει. Ευχαριστώ πολύ να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο γιατί ήταν μακρά η συζήτηση με πολύ ενδιαφέρον. Διαβάσαμε την εκτίση της κυρία Ζόμερ. Και θα αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Το πρώτο για το βενάγνωστο. Το βενάγνωστο χαρακτήρα. Ελπίζουμε ότι η θέση του Κοινοβουλίου θα μπορέσει να συνάδει με αυτή τη Συμβουλίου γιατί για μας είναι σημαντικό να έχουμε μια αναφορά μετρήσιμη για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα για την αναγνωσιμότητα, για να αποφύγουμε οι διατροφικές βιομηχανίες ακολουθούν εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά στο μέλλον. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της αναγνωσιμότητας, επιμένουμε πάρα πολύ επ' αυτού το ξέρετε και θεωρούμε ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την κατανόηση του καταναλωτή. Και για να μην αναγράφονται πληροφορίε επί ενό μέσου που εμποδίζει την κατανόηση. Τώρα, ε, γνωρίζουμε πόσο πολύπλοκη είναι η συζήτηση για ε, την προέλευση, παραδείγματος χάρη τα ψάρια φέρουν ήδη την, ε, τη σήμανση αυτή, τα λαχανικά και τα φρούτα, τα αυγά ε, φέρουν τη σήμανση για την προέλευση. Θα πρέπει να υπάρχει νομική συνέπεια μεταξύ των διάφορων διατάξεων που περιλαμβάνονται στον νέο κανονισμό. Είδατε τη θέση του Συμβουλίου για το κρέας και υπάρχουν ε, μελέτες σκοπιμότητες για τα άλλα προϊόντα, προτείνονται μάλλον μελέτες σκοπιμότητες. Ε, αυτό είναι ευθύνη της ε, ΔΕΛΤΑ Γεωργίας και της ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ, αλλά είναι σημαντικό να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες αντικτύπου πριν να σας προτείνουμε σήμανση για την χώρα προέλευσης για τα προϊόντα για τα οποία σήμερα δεν υπάρχει. Για τα αλκοολούχα αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ορισμού των λεγόμενων αλκοπόψ και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να αποσαφηνίσουμε αυτόν τον ορισμό καθώς είναι αρκετά οριστός αυτή τη στιγμή. Αλλά θα θέλαμε ο καταναλωτής να ενημερώνεται για τη σύσταση αυτών των ε, ποτών που είναι είτε αλκοολούχα είτε μη αλκοολούχα. Τώρα για τα λεργεγόνα, δεν θα σας εκπλήξω το θεωρούμε θεμελιώδες ε, να αναγράφονται αυτές οι λεργεγόνες ουσίες ακόμη και στα μη προσκευασμένα προϊόντα. Είναι σημαντικό για πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των Ευρωπαίων πολιτών που εμφανίζουν αλλεργίες. Και θα θέλουμε να διατηρηθεί η σήμανση των αλλεργιογόνων ακόμη και στα μη συσκευασμένα προϊόντα. Και θα θέλαμε να το δούμε φυσικά και στα συσκευασμένα προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τώρα την σήμανση για τα θρεπτικά συστατικά, Θεωρούμε ότι η σήμανση για τα 5 ή 6 θρεπτικά συστατικά θα πρέπει να βρίσκεται στην προστινή όψη της συσκευασία είναι προκειμένου ο τη στη στιγμή της αγοράς των προϊόντων αυτών να μπορεί να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, τις ουσιαστικές πληροφορίες για τη θρεπτική αξία. Και θα θέλαμε αυτό να διατηρηθεί στην προστινή όψη της συσκευασία για τη συζήτηση για τις μερίδες, τα 100 μιλιλίτρια, τα 100 γραμμάρια. Θα θέλαμε η σήμανση φυσικά να μπορεί να ενημερώνει τον καταναλωτή, να μπορεί να χρησιμοποιείται τη στιγμή της αγοράς ε, για να γίνονται συγκρίσεις όταν ε, συγκρίνει ο καταναλωτής ε, παρόμοια προϊόντα σε ένα ράφι του σούπερ μάρκετ, το χάρη, να μπορεί να συγκρίνει τα διάφορα προϊόντα. Και για τον λόγο αυτό προτιμούμε τα 100 γραμμάρια, τα 100 μιλιλίτρα, γιατί η σύγκριση γίνεται αμέσως και με εύκολο τρόπο. Το πρόβλημα της μερίδας, και καταλαβαίνω, αναφέρθηκα τώρα στα μπισκότα, είναι χρήσιμη τη στιγμή της κατανάλωσης του προϊόντος αυτός, Όμως για τη σύγκριση, τη στιγμή της αγοράς, θεωρούμε ότι τα 100 γραμμάρια μιλιλίτρια είναι πολύ πιο χρήσιμα για να μπορεί να επιλέξει ο καταναλωτής. Χωρίς να επιμηκύνω τη συζήτηση, αυτές είναι οι θέσει μας για τα πιο σημαντικά σημεία. Σα ευχαριστώ για το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Συγητρία. Ευχαριστώ θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχήν για τα GDA, την ημερήσια κατανάλωση, ημερήσια δόση, συστηνόμενη ημερήσια δόση. Ναι, ενδεχομένως μπορούν να προσθεθούν και νομίζω ότι εδώ συμφωνεί το Συμβούλιο. Γιατί όχι, αυτή είναι η απόφαση του Συμβουλίου. Προαιρετική όμως αναγραφή. Τώρα, τα προϊόντα που λείπουν, τα συστατικά που λείπουν. Ναι, αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για κάποια προϊόντα όπως ε, το βούτυρο παραδείγματος χάρη. Ε, όσον αφορά το κρέας θα πρέπει να δούμε γιατί το θέμα της απόψυξης παραδείγματος χάρη στο κρέας ή στο βούτυρο όντως είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν είναι όμως λάθος αυτό που ακούσαμε ότι υπάρχουν κάποια κατεψυγμένα προϊόντα τα οποία είναι τόσο πολύ ε, σύνθετα αν θέλετε που για να βάλουμε ας πούμε την ημερομηνία κατάψυξης αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές ημερομηνίες κατάψυξης. Είπατε επίσης ότι για τα συσκευασμένα και τα μη συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να αναγράφονται κάποιες πληροφορίες για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα. Βεβαίως η θέση παραμένει η ίδια. Η ημερομηνία λήξης επίσης. Ε, τα προϊόντα, παραδείγματος χάρη, που έχουν συσκευαστεί και είναι της ημέρας, φρέσκα. Η ημερομηνία θα πρέπει βεβαίως να αναγράφεται. Αλλά θα πρέπει για τα άλλα προϊόντα, τα μη προσκευασμένα, να μπορεί να δοθούν. Παραδείγματο χάνει για τις αλλεργίες. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το θέμα της συστηματικής παρακολούθησης της εφαρμογής ε, αυτής της οδηγίας. Βεβαίως. Οι πληροφορίες για την δυνατότητα να προκληθεί μια αλλεργία. Ναι, για τα συσκευασμένα προϊόντα δεν υπάρχει αμφιβολία, πρέπει να αναγράφονται αυτά τα στοιχεία με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο για τα αλλεργογόνα. Τώρα, οι μερίδες ή τα 100 γραμμάρια ή μιλιλίτρ. Το Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει ότι τα 100 γραμμάρια μιλιλίτ θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αναγραφή, όντως για λόγους συγκρισιμότητας διαφορετικών προϊόντων την ώρα της αγοράς. Και όσον αφορά τις μερίδες, πολλές φορές υπάρχουν εδώ αντιστάσεις, πολλοί θεωρούν ότι φτάνει το ότι Παραδείγματος για κάποια γλυκίσματα υπάρχει η ένδειξη ανά 100 γραμμάρια. Όντως είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ παρόμοιων προϊόντων τη στιγμή που ο καταναλωτής ε, αγοράζει το προϊόν. Γι' αυτό και επιμένουμε για τα 100 γραμμάρια ή μιλιλίτρ. Το θέμα τώρα της ένδειξης αναμερίδα, ανακομμάτι, ναι, και αυτό θα πρέπει να μπορεί να συμβεί. Και βεβαίως το θέμα της ε, ε, ημερήσιας ε, συστηνόμενης ποσότητας ή δόσης, εκεί υπάρχει θέμα με τις μερίδες. Μπορεί κανείς να, να φάει, παραδείγματος χάρη, μισό κέικ. Πώς μπορεί να καθοριστεί η μερίδα. Και σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα 100 γραμμάρια, αλλά να προσθεθεί σε αυτό την αξία ανά 100 γραμμάρια. Τώρα, η απουσία μια ουσία όπως το γλουτένιο. Εδώ, η γλουτένη, συγγνώμη. Εδώ ζητάμε εμείς να υπάρξει ένδειξη αναγραφή για κάποιο προϊόν που λείπει. Παραδείγματος χάρη στο κρασί δεν υπάρχει λίπος. Ε, ναι, εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Στην πρώτη ανάγνωση αυτή την απόφαση είχαμε πάρει. Τι άλλο ήθελα να πω. Τροπολογία 82. Ναι, εδώ ήταν η δυνατότητα που είχε προτείνει το Συμβούλιο τα κράτη-μέλη από μόνοι τους να υποχρεώσουν τους παραγωγούς να αναγράψουν το κράτος προέλευσης. Εγώ είχα πει ε, ότι εδώ είναι πιο αυστηρή και από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και το είχαμε απορρίψει. Τα κράτη-μέλη, αν θέσουν τέτοια υποχρέωση, αυτό αποτελεί εμπόδιο στις ε, ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές, το ελεύθερο εμπόριο. Γι' αυτό και είχαμε πει ότι είναι πολύ δεσμευτικό. Τώρα, η παραπλάνηση σε σχέση με τη χώρα προέλευσης. Ναι. Η σημερινή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε παραπληνητική πληροφόρηση. Στο άρθρο 7 ρυθμίζουμε όμως αυτό το θέμα της παραπλανητικής ενημέρωσης για την χώρα προέλευσης. Εμένα ξέρετε τη θέση μου για την χώρα προέλευσης. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν όμως πολλά προϊόντα που έχουν ε, ρυθμιστεί με κλαδικές, ε, τομεακές ρυθμίσεις. Και εδώ η απόφαση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση ήταν όντως λίγο ασαφής. Είχαμε πει ναι για τη χώρα προέλευσης, αλλά με μία αξιολόγηση του αντικτύπου. Ήταν όμως αυτό ο καθήκον της Επιτροπής. Εκείνη πρέπει να κάνει την αξιολόγηση αντικτύπου. Και η συνάδελφος Ροτ Μπέρεντ με παρέπεμψε στην πρώτη ανάγνωση. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου είπε, γιατί από τη μία μου λέει να επανέλθω στο αρχικό κείμενο, από την άλλη προσπαθεί να επηρεάσει το κείμενο. Παραδείγματος χάρη στην πρώτη ανάγνωση είχαμε πει ότι τα υνοπνευματόδη δεν εμπίπτουν σε, την, σε αυτό το κείμενο και τελικά βλέπουμε ότι τα alcopops προσπαθούμε να τα ξαναβάλουμε. Τα αλκοπόψ όμως, όπως ξέρετε, έχουν ένα άλλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει σήμερα σαφής ορισμός. Η Επιτροπή θα πρέπει πρώτα να βρει έναν ορισμό, Το χρειαζόμαστε, γιατί πώς μπορούμε να πάρουμε απόφαση για τα αλκοπόψ ε, αλλιώς. Και δεν συζητούμε εδώ για απλή ενημέρωση, αλλά για τις ε, θρεπτικές, για τις ενδείξεις θρεπτικών ε, τιμών. Γι' αυτό και πραγματικά τα ενοπνευματώδη είναι εκτός. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Αν όμως ξαναδώσω το λόγο σε διάφορους ομιλητές, μετά θα πρέπει να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Οπότε δεν τελειώνω με τίποτα. Είμαι στα χέρια σας, κάνω ό,τι θέλετε ένα σημείο μόνο. Εσείς και η κυρία Γκαρδίνη ένα σημείο. Εντάξει, κυρία Βιγμούτ. Ένα μικρό σημείο, κυρία Σόμερς. Δεν μπορείτε να επιλέγετε ποια από τις θέσεις του Κοινοβουλίου θα κρατήσετε. Συμφωνώ για το ενόπνευμα. Το χάσαμε το επιχείρημα εκεί. Αλλά κερδίσαμε το, το, το επιχείρημα για την εμπρόστια όψη. Πέντε συστατικά και για τη χώρα προέλευση. Δεν μπορούμε να λέτε ότι δεν θα ε, υποστήσετε τη θέση του Κοινοβουλίου για τους, ε, τα πέντε στατικά μπροστά στο πακέτο. Διερωτώ με τελικά θα δεχτείτε την ε, κοινή θέση του Κοινοβουλίου, τη θέση του Κοινοβουλίου μας πρώτη ανάγνωση. Ε, τελικά δεν είναι αυτό όμως που υποστηρίζετε, έτσι, εδώ. Κυρία Γκαρντίνη, ένα ερώτημα. Λέτε ότι δεν μπορεί να γράφει, δεν περιλαμβάνει ε, γλουτένη. Ε, η γλουτένη είναι μια ουσία που πολλά άτομα είναι αλλεργικά. Είναι σημαντικό να βάζουμε επίσης ότι δεν, περιλαμβάνει, δεν περιέχει και ίχνη γλουτένης, γιατί μερικές φορές και ίχνος μπορεί να δημιουργήσει δράμα. Ε, σε αυτές τις ουσίες υπάρχουν παρεκκλήσεις. το βασικό είναι να λέμε ότι αυτές οι αλλεργικές ουσίες, να το γράφουμε, να γράφουμε ότι δεν, δεν υπάρχουν αυτές οι ουσίες. Καλύτερα να βάζουμε δύο-τρία στοιχεία παραπάνω παρά να πεθάνει κάποιος από αναφυλακτικό σοκ. Υπάρχουν και τα κεράσια. Ε, που δημιουργούν πρόβλημα. Επομένως, αυτό που είπε η καρτίνα είναι σωστό. Κυρία Σόμερ, και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ε, μπερδεύεται τα 100 γραμμάρια με τα 100 ε, μιλιλίτρ και τις μερίδες. Οι μερίδες είναι ένα τμήμα Εμείς ζητάμε οι επιχειρήσεις, αν έχουν 20 κομμάτια μέσα σε ένα πακέτο 100 ε, μιλιγκράμμ, να βάζουν να βάζουν τα γραμμάρια που ζυγίζει το κάθε τεμάχιο. Έτσι, πέντε ας πούμε. Αν θέλει ας πούμε κάποιος να συγκρίνει τα 100 γραμμάρια ενός προϊόντος που παράγεται από μια εταιρεία με τα 100 γραμμάρια ενός προϊόντος που παράγεται από άλλη εταιρεία, οκ. Αλλά γιατί να αποκλείσετε τη δυνατότητα να ξέρουμε κάθε μερίδα που είναι μικρότερη από τα 100 γραμμάρια τι περιλαμβάνει. Γιατί. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή και θέλω να το εξηγήσετε, κυρίω ε, κομισιόν. Θέλετε, θέλετε να προστατεύσετε όλη την Ευρώπη. Καλό να την προστατεύσετε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο την επιχείρηση που παράγει κάτι, κυρία Ρουτ Μπέρεν, πολύ σύντομα και μετά η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Είναι θεσμικό το θέμα. Όλοι ξέρουμε ότι στη δεύτερη ανάγνωση δεν μπορεί κανείς να προσθέσει κάτι που δεν έγινε δεκτό στην πρώτη ανάγνωση. Μα γι' αυτό και είναι άχρηστη συζήτηση για τα αλκοολούχα ποτά. Το ξέρουμε αυτό. Στην πρώτη ανάγνωση εμείς σε καμία, μα σε καμία περίπτωση δεν μιλήσαμε για εθελοντικό χαρακτήρα όσον αφορά τα 100 γραμμάρια, τα 100 μιλιλίτ και τις μερίδες. Είπαμε υποχρεωτικά Υποχρεωτικά. Δεν είπαμε επίσης ότι είναι ε, προαιρετική η αναγραφή της χώρας προέλευσης. Εμείς μιλήσαμε στους 28 για υποχρέωση. Και αυτά έπρεπε να είναι στη δεύτερη ανάγνωση. Κυρία Σόμερ. Νομίζω πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Νομίζω ότι για τη γλουτένη υπάρχει μια παρανόηση. Δεν μιλήσαμε εμείς για αυτήν την ουσία. Για τις, αλλεργι... για τις αλλεργογόνες ουσίες σαφώς και θα υπάρχει ένδειξη. Εγώ μίλησα για το άρθρο 7, για παραπλανητικές πληροφορίες όσον αφορά άλλες ουσίες, όχι αυτές που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης για τη χώρα προέλευσης ήταν ασαφής. Αν διαβάσετε καλά την έκθεσή μου θα το καταλάβετε αυτό, θα το διαπιστώσετε. Επίσης, το τι θα αναγράφεται στην πρώτη, ε, μάλλον στην προστινή όψη του πακέτου, είχαμε ένα σαφέστατο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Οχτώ ή εννέα ουσίες συστατικά. Άλλοι είπαν όμως ότι έγινε λάθος και δεν μας αρέσει αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν, κοιτάξτε την τροπολογία 1. Για όλα αυτά που αποφασίσαμε στην πρώτη ανάγνωση, αν δεν θεωρείτε ότι αντικατοπτρίζονται οι θέσεις σας στη δεύτερη. Και κυρία Ροτ Μπέρεντ, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι εσείς εδώ κάνετε μια συζήτηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ τα μέσα στη Γερμανία και όχι την Ευρώπη. Είναι προσωπική η επίθεση που μου κάνετε και τη θεωρώ υπερβολική. Πραγματικά νομίζω ότι πρέπει εδώ να ακολουθήσουμε την κανονική και ομαλή διαδικασία. Συνήθως δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον τόνο στο Κοινοβούλιο. Συνήθως ε, είμαστε ευγενεί και καλό θα είναι να παραμείνουμε ευγενεί. Υπενθυμίζω, η 18 Μαρτίου είναι η κατάθεση των τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι, στις 12, ψηφίζουμε, 12 ε, Απριλίου ψηφίζουμε ε, στην Επιτροπή